Bueno, Θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Εν συντομία. Θα κάνω δύο-τρεις ανακοινώσεις από πλευράς Προεδρίας τις οποίες δεν μπόρεσα να κάνω σήμερα το πρωί, θέλω καταρχάς να δηλώσω απερίφραστα ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως και ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μογκερίνη, για την παρουσία της στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα, γιατί καταφέραμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα πολύ καλό νέο για όλους εμάς οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είδαμε τη δέσμευση της κυρίας Μογκερίνη η οποία εξέφρασε τη βούλησή της να είναι ενεργή σε αυτό το πεδίο εξ αρχής στην πρώτη ολομέλεια του νέου έτους. Έχουμε υιοθετήσει διάφορα ψηφίσματα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, την περίπτωση του Αλεξέη Ναβάλνη στη Ρωσία, την περίπτωση του Πακιστάν και την κατάσταση μετά την επίθεση στο σχολείο της Πεσαβάρ. Επίσης εξετάσαμε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος το θέμα της Αιγύπτου και παράλληλα συντάξαμε μια επιστολή. Αυτή είναι μια δράση, ξέρετε, που, στην οποία καταφεύγουμε όλο και πιο συχνά. Συντάξαμε λοιπόν μία επιστολή στο πρέσβη του βασιλείου του Μπαχρέιν για την κράτηση του Σεΐχη Αλίξ Ακμάνε που αποτελεί ε, μέλος ε, της ε, αντιπολίτευσης της ομάδας αυτής. Παρακολουθήσαμε την ε, σύγκρουση στο Μπαχρέιν και θα ε, παρακολουθούμε εκ του σύνοικης τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο. Σε γενικές γραμμές ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει βρει τη θέση του στην Ολομέλεια και θα πρέπει αυτό το χώρο, αυτό το διάστημα ε, που έχουμε στην Ολομέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα να το διατηρήσουμε οπωσδήποτε. Σίγουρα πρέπει να το βελτιώσουμε, αλλά είναι κίνητρο για να ε, συνεχίζουμε να αφυπνίζουμε τις συνειδήσεις και να έχουμε καλύτερη αγωγή του πολίτη όλοι μας. Έχουμε υιοθετήσει σχετικά κείμενα για το νόμο που απαγορεύει την προπαγάνδα στο ε, Κυργυζία σε σχέση με τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, μια κείμενο το οποίο καταφέρεται εναντίον βεβαίως αυτού του νόμου. Έχουμε ε, και τον, ε, την περίπτωση Ραΐφ Μπαντάουι στη Σαουδική Αραβία, για την οποία θα μιλήσουμε και αργότερα, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο σε χίλιες βουρδουλές, τις οποίες θα υποστεί σε βάθος διαφόρων μηνών, αρκετών μηρών μηνών και αυτή την Παρασκευή θα μαστιγωθεί ε, για να εκτίσει μέρος της ε, ποινής του. Θα ανταλλάξουμε απόψεις για αυτή την κατάσταση και ε, θα ακούσουμε μαρτυρίες από τη σύζυγο και την κόρη του. Προχωρούν λοιπόν τα πιο σοβαρά περιστατικά, τα πιο σοβαρά ζητήματα, δεν τα αφήνουμε. Έχουμε και την περίπτωση της Λέιλα Γιούνου και θα προσεγγίσουμε και αυτή την περίπτωση αργότερα. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι τα πιο επίγοντα τα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και δεν τα παραγνωρίζουμε. Ερχόμαστε τώρα στις ερωτήσεις. Ο συνάδελφος που προτείνει την ερώτηση πρέπει να τη διατυπώσει μέσα σε δύο λεπτά, σε λίγο χρόνο, έτσι ώστε αυτοί που θα πρέπει να απαντήσουν, δηλαδή οι υπεύθυνοι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την εξωτερική δράση, να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Ξεκινούμε λοιπόν με την ερώτηση του κυρίου Ντεβεσμάκερ για την κατάσταση των κοριτσιών στο Τσίβοκ που απήχθησαν από την οργάνωση Μπόκο Χαράμ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να θέσετε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η Μποκο Χαράμ συζητιέται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η Μποκο Χαράμ γίνεται όλο και πιο βίαιη, πιο ε, βάρβαρη και υπάρχουν πάρα πολλά επίθετα που θα μπορούσα να παραθέσω. Πάντως εκείνο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε όλο και περισσότερα φαινόμενα μαζικών εκτελέσεων. Η Μποκοχαράμ αρχίζει να παρισφρέει και σε γειτονικές χώρες και θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Καταρχήν, όσον αφορά τα κορίτσια του Τσίμποκ ε, του σχολείου, απηχθήσαν ε, από την Χαράμ, πάνω από 200 κορίτσια και πολλά εξ αυτών εξακολουθούν να παραμένουν στα χέρια της Χαράμ. Ακόμα και μία μέρα το να βρίσκεται κανείς εχμάλωτος είναι πάρα πολύ, αλλά εννέα μήνες είναι υπερβολικά πολύ. Εξάλλου πάρα πολλά από αυτά τα κορίτσια βιάστηκαν, ορισμένα εξ αυτών επανειλημμένα και ορισμένα πάλι εξ αυτών βρίσκονται στην ε, τελική φάση της εγκυμοσύνης. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουν τις αρχές της Νιγηρίας να προχωρήσουν στην ε, απελευθέρωση αυτών των κοριτσιών. Μήπως λοιπόν μπορείτε να μας ενημερώσετε λιγάκι ή να μας πείτε εν πάση περιπτώσει κατά πόσον έχετε σημειωθεί κάποια, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Δεύτερον, η ε, τελευταία επίθεση στην Κάμπα. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Πρόκειται για ένα καταβλισμό με 102.000 με πάρα πολλούς ε, πρόσφυγες και ε, εκείνο που είναι σαφές είναι τελικά ότι η Μπόκο Χαράμ αποκτά όλο και μεγαλύτερη εξουσία, γίνεται επαρμένη. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια διεθνή στρατηγική για να αντιμετωπίσει την, ε, αποτελεσματικά την ε, τρομοκρατία και διαρωτώ με τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Θα έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι ένα θέμα που συζητήσαμε με την κυρία Μογκερίνη την περασμένη Τετάρτη. Ε, ποιος θα απαντήσει Good afternoon. Thank you for inviting me to this question time on Nigeria. Dr. I'm in charge. Ε, Καλησπέρα, λέγομαι Βαλχάιμ, Dr. Βαλχάιμ, ασχολούμαι με τα θέματα της Νιγηρίας. Θυμόσαστε όταν απήχθησαν στο Τσίμπουκ τον Απρίλιο τα κορίτσια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσα καταδίκασε την απαγωγή και είπα τους εκπρόσωπος στις 17 Απριλίου εξέδωσε δήλωση εκφράζοντας αλληλεγγύη και ζητώντας άμεση απελευθέρωση των κοριτσιών και υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, ζήτησε. Έκτοτε προφανώς υπήρξαν πολλές δηλώσεις, πολλοί διάλογοι και όπως είπα την περασμένη εβδομάδα έγινε πλήρη συζήτηση στην Ολομέλεια. Η κυρία Μογκερίνη εκεί απάντησε στις τεθήσεις ερωτήσεις. Η κρίση της ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων και των απαγωγών των κοριτσιών προφανώς έχει μεγάλη προτεραιότητα στο διάλογο με την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Συζητήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, στο διπλωματικό διάλογο που έγινε 27 Νοεμβρίου στην Αμπούτζα. Σε αυτό το διάλογο η Ένωση ζήτησε από την κυβέρνηση της Νιγηρίας να αυξήσει τις προσπάθειες που καταβάλει. Όχι μόνο για να ελευθερώσει και να επιστραφούν τα κορίτσια, αλλά να εκριζώσει τις βιο... τη βία και να σταματήσουν οι απαγωγές. Επανειλημμένα στείλαμε μήνυμα στις Νιγηριανές αρχές λέγοντας ότι πρέπει να θετήσουν σφαιρική προσέγγιση. Όχι μόνο στα στατιωτικά μέτρα, αλλά να εκριζωθούν και τα αίτια της βίας. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στην προστασία του πληθυσμού, κυρίως των γυναικών και των παιδιών. Οι καρδιές και τα μυαλά και το πνεύμα των ε, ανθρώπων πρέπει να είναι ένα κατά της Μποκοχαράμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά από τις δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας. Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις προσπάθειες της Νιγηρίας με διάφορες παρεμβάσεις. Έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιτρομοκρατικό που έχει δρομολογηθεί στο μέσο που συμβάλλει σταθερότητα και την ειρήνη. Βοηθά την ε, αύξηση δυναμικού της υπηρεσίας ε, του Συμβούλου Εθνική Ασφάλεια σε θέματα αντιτρομοκρατία, ε, να, ε, να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην υπάρχουν ριζοσπαστικέ ε, θέσει και ο ποινικό τομέα, ο ποινικό κώδικα να διαμορφωθεί και 10 εκατομμύρια θα δοθούν ούτω ώστε να βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην ασφάλεια και στην ειρήνη και η συμμετοχή του και υπάρχει και συνιστόσα που αφορά τι γυναίκε, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, συνιστόσα για την πρόσβαση σε προστασία και ε, συστήματα καταγγελιών για τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπόκεινται σε φαινόμενα βίας λόγω φύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτησε πρόσφατα μια απόφαση για ένα πρόγραμμα με τη UNICEF που έχει σαν στόχο την αύξηση της προστασίας που παρέχεται ε, και να βελτιωθεί όλη η κατάσταση παιδιά που ζουν ε, στις περιοχές που είναι υπό μουσουλμανικό έλεγχο και που είναι και το τσίμπο και έχει κηρυχθεί κατάσταση ανάγκης. Τα παιδιά που έχουν πληγεί θα τύχουν ψυχολογική στήριξη. Και ξεκίνησε το μέτρο τον Ιανουάριο. Η Νιγηρία είναι με στήριξη όσον αφορά και την εταιρική σχέση για την παιδεία και συμβάλλουμε εμεί χρηματοδοτικά σε αυτό το πλαίσιο. Μετά τι απαγωγέ του Τσίμποκ, τα κράτη μέσα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω άφησαν την υποστήριξή τη προ την Νιγηριανή κυβέρνηση. Κάποια κράτη ε, διέθεσαν και βοήθεια όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών, ε, επιχειρήσει κατά των παγωγών και ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση τη δυνάμει ασφαλεία στην Ιγυρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια κράτη-μέλη επίση ενεργά συμμετέχουν στι διασκέψει για περιφερειακή ασφάλεια που έχουν διεξαχθεί από το Μάιο 2014 έκτοτε. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε το Μάιο, η δεύτερη στο Λονδίνο τον Ιούνιο, η τρίτη στην Αμπούτζα το Σεπτέμβριο και χτε μόλι έγινε και τέταρτη διάσκεψη για την ασφάλεια στην Ιάμι. Αυτές οι διασκέψεις ασφαλείας ε, συναθρίζουν την Ιγυρία και τις γειτονικέ χώρες και διεθνείς εταίρους και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα εκπροσωπεί το σε επίπεδο. Χθε ήταν ειδικό εκπρόσωπος για τη Σαχέλ παρόν. Ε, στο διάλογο στις διασκέψεις αυτές επανειλημμένα έχουμε τονίσει την ανάγκη που υπάρχει για ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία και έχουμε ζητήσει επιτάχυνση της εφαρμογής ε, των δεσμεύσεων που έχουν αληθεί από τις διασκέψεις. Να δημιουργηθεί πολυεθνική ομάδα κρούσης να γίνονται κοινοί ε, μεθοριακοί έλεγχοι ε, και να υπάρχει και ένα κέντρο συλλογή των πληροφοριών των μυστικών περιοχών τη περιοχή. Μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ιγυρία και τι γειτονικέ χώρε στην καταπολέμηση τη δημοκρατία. Περιέγραψε ήδη κάποιε δραστηριότητε που έχουν δρομολογηθεί. Εν τέλει όμω, μόνο με ισχυρή περιφερειακή συνεργασία και περιφερειακή ηγεσία, όπου η Νιγηρία θα ηγείται, Μόνο τότε θα μπορεί να ξεπεραστεί ο κίνδυνος και η απειλή. Όπως είπατε, η τρομοκρατία έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκή Ενώσεως, όχι μόνο τώρα, αλλά εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Βασικά θέματα, ένα από τα βασικά θέματα του Συμβουλίου της 19 η Ιανουαρίου, ε, εξωτερικών υποθέσεων, τα τρομοκρατία. Και το Φεβράριο θα συζητηθεί η Αφρική, ε, και οι ριζοσπαστικέ θέσει και η τρομοκρατία σε αυτή την ε, Ήπειρο, την Αφρικανική Ήπειρο, θα συζητηθούν. Εν ώψη αυτών, οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω αναλύουν το πώ περαιτέρω θα αυξήσουμε την υποστήριξη που παρέχουμε και ρωτήσατε ε, ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, σαν ανταπόκριση της απειλής από πλευράς Μποκοχαράμ. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τις λεπτομέρειες της στρατηγικής που έχει δρομολογηθεί, αλλά να τη ρυθμίσουμε ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις. Και στόχο στόχος θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, η οποία σημαίνει καθημερινά και βέβαια να συγκρατηθεί η απειλή, ξεκινώντας από την προστασία ε, των, ε, ε, πληθυσμών, γυναίκες και παιδιά. Θέλουμε να στηρίξουμε κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες που θα δημιουργηθούν, να παρέχονται βασικές υπηρεσίες και θέλουμε να υπάρξει δυνατότητα αντοχής του πληθυσμού στις δοκιμασίες. Και θέλουμε να υπάρχει λογοδοσία όσον αφορά τα θεσμικά όργανα που κινούνται και λειτουργούν. Θέλουμε να αυξηθεί η περιφερειακή συνεργασία για να ξεπεραστούν τα άμεσα προβλήματα ασφαλείας, αλλά θέλουμε και μακροπρόθεσμα να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή και συζητάμε με όλες οι πιεστές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΚΟ, ε, εκπροσώπους του μέσου και την εξωτερική πολιτική και άλλους φορείς, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε δεόντως τις πολιτικές μας. Όταν είπα ότι συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Όπω το δυτικό προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με συναδέλφου για τη διαχείριση των κρίσεων και το σχετικό σχεδιασμό. Σε αυτού αναφερόμουν. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεμέσ Μέικερ είναι ικανοποιημένο με την απάντηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, όμως θα ήθελα να θέσω ε, να, να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κορίτσια. Ε, έχουμε, ξέρουμε ποιες πρωτοβουλίες έχουν δρομολογηθεί, ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την εκρίζωση του προβλήματος. Αυτό είναι καλό. Συγκεκριμένα όμως, έχουμε 200 κορίτσια που πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως, το ταχύτερο δυνατόν. Υπάρχει κάποια πρόοδος όσον αφορά αυτή την πτυχή του προβλήματος. Ξέρω ότι σε κάποιο βαθμό είμαστε και αδύναμοι, ανίσχυροι αλλά τίθεται το ερώτημα, έχουμε και κάποια θετικά μαντάτα. Και μια άλλη ερώτηση για την επίθεση στην Πάργα. Η αντιπροσωπεία μας στην Αμπότζα ε, συμμετέχει στην προσπάθεια εξευρέσεως των ε, αιτίων. Κοιτάξτε, όσον αφορά την απαγωγή των κοριτσιών, όπως και εσείς και εμείς έχουμε υποβάλει αυτή την ερώτηση στις συζητήσεις που είχαμε με τις αρχές της Νιγηρίας. Τις ρωτήσαμε αν έχουν κάποια νέα από τα κορίτσια και είπαν όχι. Γνωρίζουν ότι τα κορίτσια κατά πάσα πιθανότητα έχουν μοιραστεί σε διάφορους καταπλησμούς, δεν είναι όλα μαζί πλέον και παρά τις πληροφορίες που έχουν δώσει κάποια από τα κράτη-μέλη τα οποία μάλιστα επέβαλαν και κάποια σχέδια για ε, πτήσεις πάνω από την περιοχή και είχαν και κάποια σχέδια για συγκεκριμένες επιχειρήσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προκλήσεις παρά λοιπόν αυτή την υποστήριξη τελικά δεν μπορούμε να πούμε ότι σημειώθηκε πρόοδος δυστυχώς ε, τον Νοέμβρη στην τελευταία συνάντηση κάναμε την ίδια ερώτηση και οι Υπουργοί Εξωτερικών δεν είχαν καμία συγκεκριμένη απάντηση. Ε, τώρα, ο διάλογος με τους αρμόδιους στην Ιγυρία για την ασφάλεια και την άμυνα ε, δεν είναι εύκολος. Ε, Μπλέκονται διάφορες υπηρεσίες και δεν είναι και πάντα τέλεια και καλά συντονισμένες άρα δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς μαζί τους και να αποκομίσει τις καλές σωστές απαντήσεις. ξέρετε ότι στην Ιγυρία ε, δεν υπάρχει ε, εκπροσώπηση δική μας, ε, δεν υπάρχει σύμβολος ασφαλείας στη χώρα και ως εκ τούτου ο διάλογος γίνεται πολύ δύσκολος διότι δεν έχουμε το σωστό συνομιλητή για να μπορούμε να μιλήσουμε με τους αρμόδιους ασφαλείας στην Ιγυρία. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, αυτή είναι η στρατηγική μας για να βελτιώσουμε τη δυνατότητά μας για θέματα ασφαλείας. Τα κράτη-μέλη που έχουν αυτή τη δυνατότητα ε, δεν ε, προσφέρουν ε, εύκολα τουλάχιστον πληροφορίες για τέτοιου είδους θέματα. ενημερώνουν κάπως ε, και όσον αφορά τα κορίτσια δυστυχώς δεν έχουν πληροφορίες. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Όσον αφορά την επίθεση στην Μπάγκα γνωρίζετε ότι ξεκίνησε με την κατάληψη της στρατιωτικής βάσης στην Μπάγκα. Η Μπάγκα είναι ο χώρος όπου υποτίθεται θα ε, είχε τη βάση της η Task Force. Ε, εκεί όμως ε, υπάρχουν μόνο ε, νιγηριανές δυνάμεις γιατί οι άλλες χώρες αρνήθηκαν να στείλουν δυνάμεις τους λέγοντας ότι η μπάγκα είναι πολύ επικίνδυνη ως βάση για να εστιαστεί το χώρο αυτό η πολυεθνική δύναμη. Μετά από λίγε μέρες η Μπόκο Χαράμ επιτέθηκε όχι μόνο στην Μπάγκα αλλά και στα 16 γειτονικά χωριά. Ε, σκοτώθηκαν από 200 μέχρι 2.000 ε, πρόσφυγες, εκτοπιστέντες και πάλι ε, είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς τις σωστές πληροφορίες. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε ίσως επιβεβαίωση των αριθμών αυτών, αλλά... δεν πιστεύουμε ότι είναι τελικά 2.000 άτομα, κατοντάδες πρέπει να είναι, πολλοί είναι φυσικά και αυτοί, αλλά δεν μπορούμε να σας πούμε με απόλυτη ακρίβεια ακρίβεια πόσοι δολοφονήθηκαν. Ε, επίσης ε, ε, δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε ακριβώς γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτή την περιοχή. Χιλιάδες προσφύγων κατέφυγαν στις όμορες χώρες. Εμείς παρακολουθούμε εκ του σύνεγης όλες αυτές τις εξελίξεις. Αποκινούμε τα κράτη-μέλη, παρακολουθούμε την κατάσταση και όπως σας είπα έχουμε διάλογο με την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Το θέμα θα είναι πρώτη προτεραιότητα και στις συζητήσεις ε, που θα ακολουθήσουν. Τώρα προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε τη στρατηγική μας για να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση της απειλής της Μποκοχαράμ που αφορά όχι μόνο την Ιγυρία αλλά και τις γειτονικές χώρες και τελικά όλους μας. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια στρατηγική που θα δείχνει ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λογικά δεν θα πρέπει να υπάρχουν ερωτήσεις ή τελειώς δεν θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Όμως θεωρώ ότι το δεύτερο μέρος της απάντησης είναι πραγματικά απάντηση στην ερώτηση που είχε θέσει ο κύριος Ντεπνισμέκερ. Ε, σας παρακαλώ να είστε συγκεκριμένοι στις ερωτήσεις γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις και λίγο χρόνο. Επομένως να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις και να δίνετε και συγκεκριμένες απαντήσεις. Ε, επόμενη μελήτρια για το θέμα του Νεπάλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε για την Επιτροπή Εκεχηρίας και Συμφωλίωσης το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, ε, είπα τη αρμοστία, ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ ε, άσκησαν κριτική ε, και είπαν ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι επαρκές, ε, <coughs> δεν πληρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, διότι π.χ. επιτρέπει αμνηστία για αδικήματα τα οποία τιμωρούνται βάσει του διεθνούς δικαίου. Δεν έγινε δήλωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με μια φωνή για το θέμα αυτό ούτε εξέδωσε δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έγκριση αυτού του νομοσχεδίου. Ε, και επομένω, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερω για το κράτο δικαίου και το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί δεν εξέδωσε δήλωση για να ενθαρρύνει πρωτοβουλίε που θα αποδώσουν δικαιοσύνη και για να αποτρέψει αυτού που θα απομακρύνουν του εγκληματίε από το να έχουν ατιμορρησία. Στη συνέχεια, Πώς γίνεται η παρακολούθηση όλων αυτών. Στη, δίδεται στήριξη στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τα προβλήματα που έχουν σχέση με το νόμο αυτό, π.χ. δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα των θυμάτων σε αποζημίωση. Ε, μειώνεται η δυνατότητα της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη συμφιλίωση έτσι τίθεται αναμφιβόλο η ακαιρεότητα των υποθέσεων των φακέλων που είναι στο δικαστικό σύστημα. Ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά. Και τελευταίο ερώτημα που δεν έχει σχέση με αυτό το νόμο αλλά με ένα άλλο στοιχείο το οποίο φάνηκε στο βιβλίο του Τόμας Πέλινγκ τον Αύγουστο του 2014 περιγράφει την ευρωπαϊκή συνεργασία σε μαζικές καταστρατηγήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Νεπάλ. Η MI6, η ΜΙΙΟΤΑ6 εκπαίδευσε ε, ε, στρατιώτες στην επιχείρηση Mustang, κάτι το οποίο οδήγησε και σε συλλήψεις και σε ε, θανάτους. Το γνώρισε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ναι, ε, ποια ήταν η θέση της εναντί αυτών των ισχυρισμών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ο κύριος Πίτερ Νάγκη έχει το λόγο για να απαντήσει. Thank you, uh, Madam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανταλλαγή απόψεων για τον ΕΠΑΛ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ερωτήσεις. Αυτή η Επιτροπή της Αλήθειας και της Συμφιλίωσης, μάλλον ο νόμος είναι ένα σημαντικό θέμα για την όλη ε, εξομάλυνση καταστάσεως στο Νεπάλ. Δύο επιτροπές δημιουργούνται, η μία που αφορά την αλήθεια και τη συμφιλίωση και η άλλη αφορά την έρευνα των ε, εξαφανιθέντων ατόμων. Αλλά υπολείπεται των διεθνών προδιαγραφών η νομοθεσία όσον αφορά τη μεταβατική δικαιοσύνη. Και ένας αξιότιμος βουλευτής αναφέρθηκε σε αυτές τις ε, ελλείψεις και γνωρίζουμε σαν υπηρεσία εξωτερικής δράσης αυτά τα θέματα και τα θύματα και οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσέφηγαν στον το δικαστήριο του Νεπάλ κατά τη νομοθεσία. Και η κατάσταση εκκρεμεί για την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ τι εξελίξει και τη διαδικασία ειρήνευση την υποστηρίζει και το θέμα τη μεταβατική από τη δικαιοσύνη που είναι ένα σημαντικό λιθαράκι στην όλη προσπάθεια. Σε τακτικέ επαφέ με τις αρχές του Νεπάλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με νομικούς εμπειρογνώμονες ζήτησε ένα μοντέλο μεταβατικής δικαιοσύνης που θα ταιριάζει με τις διεθνείς προδιαγραφές. Και ανησυχίες για το νομοσχέδιο έχουν εκφραστεί σχετικά με όλα αυτά που συζητούμε. Σε ύψιστο πολιτικό επίπεδο θα θυμόσαστε ότι οι πρόεδρος Φαν Ρομπάι και Μπαρόσο συζήτησαν το θέμα της ειρήνης ε, με τον Πρωθυπουργό Κοϊράνα, τον Πρωθυπουργό του Νεπάλ, όταν είχε τον περασμό Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες. Και ο πρώην Επίτροπος κ. Πίμπαλξ το έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νεπάλ το μήνα Οκτώβριο, μερικές εβδομάδες αργότερα με άλλα λόγια. Ε, πιστεύουμε ότι η μέθοδος μας, δηλαδή ε, να δίνουμε παρενέσεις και να στηρίζουμε βοηθά τη μεταβατική διαδικασία στο Νεπάλ αλλά δεν έχουμε φτάσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Μια συγκεκριμένη δήλωση για το νομοσχέδιο σε αυτή τη φάση θα ήταν κάτι αντιπαραγωγικό διότι η όλη ειρηνευτική διαδικασία είναι πολύ ευαίσθητη. Περιμένουμε ένα νέο σύνταγμα του Νεπάλ που είναι στο επίκεντρο της όλης προσπάθειας ειρήνευση στο Νεπάλ. Ε, ε, έχουν θέσει την προθεσμία 22 Νοεμβρίου οι κάτοικοι του Νεπάλ, αύριο. Σίγουρα δεν θα τηρηθεί η προθεσμία. Εμεί ενθαρρύναμε την πολιτική ηγεσία να καταλήξει σε συνένεση. Εν ώψη λοιπόν των εντάσεων που υπάρχουν στο Κατμαντού, που σχετίζονται ε, με την αναμενόμενη υπέρβαση της προθεσμίας οι εκπρόσωποι μα στο Κατμαντού ε, δήλωσαν, έκαναν δήλωση εκ μέρου της διεθνούς κοινότητας στο Νεπάλ. Δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι λέει η δήλωση. Εκφράζει ανησυχίε. Και παροτρύνει όλα τα μέρη να επιστρέψουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Στηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία στο Νεπάλ οικονομικά. Μέσω του ε, Ταμείου για την Ειρήνη στο ΕΠΑΛ. Έχουμε τέσσερα προγράμματα για την απελευθέρωση θυμάτων συγκρούσεων και την αποκατάστασή τους. Ε, κυρίως εκτοπιστέντες ε, και άτομα με αναπηρία έχουμε σαν στόχο. Στηρίζουμε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολούνται με την κληρονομιά των συγκρούσεων, θέματα βασανιστήριων, εξαφανίσεων ε, και πληγέντων παιδιών. Όσον αφορά συγκεκριμένο ερώτημα, για το βιβλίο του Τόμας Μπέλ η ε, υπηρεσία εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντέδρασε όταν εξεδόθη το βιβλίο. Ήδη τον Αύγουστο υπόθηκε κάτι. Δεν ενδείκνεται να πούμε κάτι παραπάνω τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να υποστηρίζει εκ του σύνεγγυς την όλη μετάβαση στο Νεπάλ, τη συνταγματική διαδικασία. Στόχος ποιος είναι. Το Νεπάλ να ακολουθήσει μια, δημοκρατική, μια ειρηνική δημοκρατική μετάβαση σύμφωνα στι διεθνεί προδιαγραφέ. Το ίδιο ισχύει για το νομοσχέδιο. Όμω το ίδιο το Νεπάλ πρέπει να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχουμε μία ερώτηση από τη συνάδελφο κυρία Άννα Γκόμες η οποία δεν είναι εδώ, αλλά θα την αντικαταστήσω εγώ για την Αιθιοπία. Και η ερώτηση είναι η εξή. Ποιε είναι οι δράσει, ποιε είναι οι προσπάθειε που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εγγυηθεί την απελευθέρωση των, ε, του Εσκίντερ Νέγα, του Ρίγιο Ταλέμου και του Αντικανατσέφ Σέγκε. Ο τρίτος είναι Βρετανός υπήκος οι πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν βοηθήσει τους κρατούμενους, τους έχουν επισκεφθεί στη φυλακή, έχουν ελέγξει ε, ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους. Γνωρίζουμε ότι ένας από αυτούς είναι σοβαρά άρρωστος. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε βάθος χρόνου στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιθιοπίας. Νομίζω ότι η κυρία Βικτόρια Γκυγέν είναι η υπεύθυνη και αρμόδια να απαντήσει. Παρακαλώ. σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξετάσουμε τα θέματα που έχει θέξει η κυρία Γκόμες. Εγώ είμαι αρμόδια για το κέρα της Αφρικής, ε, την Ανατολική Αφρική στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έτσι για να έχουμε μια εικόνα θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυσχηδείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αιθιοπία. Θα αναφερθώ σε θέματα ανθρωπίων δικαιωμάτων, ασφάλειας και σε πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε λοιπόν ε, έναν ουσιαστικό έντονο διάλογο με τις αρχές της Αιθιοπίας στο ανώτατο επίπεδο. Και ε, στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου επανειλημμένα έχουμε επισημάνει τη σημασία των πολιτικών ελευθεριών, της ε, ελευθερίας έκφρασης, αλλά επίσης και πόσο σημαντικό είναι να αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στις δίκαιες δίκαιες στην πολιτική δικονομία. Επίσης εκφράζουμε τις ανησυχίες μας ε, για ε, τις ε, αντιτρομοκρατικές ενέργειες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει τις ανησυχίες της, κυρίως πέρυσι το έπραξε αυτό, με σχετικά με τη δημοσίευση δύο δηλώσεων που αφορούν στην σύλληψη δημοσιογράφων, blogger και μελών της αντιπολίτευσης έχουμε ε, παρακολουθήσει επιτόπου την δίκη στην Αντίσα Μπέμπα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών ε, στην Αντίσα Μπέμπα παρακολούθησαν τη δίκη των τριών ατόμων, η Ιτελέμο και Γκάτσα Τρία άτομα λοιπόν που έχουν διπλή πικότητα την ε, ε, ηθαγένεια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αιθιοπίας. Είμαστε σε στενή επαφή με τους συγγενείς και την οικογένεια των ε, προφυλακισμένων και μπορούμε να τους βοηθήσουμε οποτεδήποτε το ζητήσουν. Αυτό συνέβη ήδη το 2013 όπου ο Νταλίμ ε, αποφάσισε να κατέβει σε απεργία πείνας, ε, η οικογένειά του μας ε, πλησίασε και εμείς συμπεριλάβαμε το θέμα αυτό στις συζητήσεις μας με την κυβέρνηση. Επίσης αφορά τον κρατούμενο Τσέγγι. Το Σεπτέμβρη στην ίδια επιτροπή συζητήθηκε η υπόθεσή του. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει ανεπιφύλακτα το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει πρόσβαση ε, σε συζητήσεις με τον προφυλακισμένο. Δύο φορές έγινε αυτό και μας ενημέρωσαν ότι μέχρι και το Δεκέμβρη ήταν σε καλή κατάσταση. Ε, και κάτι άλλο που δεν μας έχει ζητηθεί αλλά θέλω να προσθέσω ότι θα γνωρίζετε κατά πάσα πιθανότητα ότι η Αιθιοπία έχει επίσης καταδικάσει δύο Βρετανούς ε, αιθιοπικής προέλευση 15 Ιανουαρίου που θέλησαν να συστήσουν Ισλαμικό κράτος στην Αιθιοπία. Και πάλι στηρίζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο επιθυμεί να έχει πρόσβαση μέσω του προξενείου ε, και να διασφαλίσει μια δίκαιη δίκη. Η ε, Αιθιοπία είναι βασικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς. Προφανώς ε, στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή η Αιθιοπία συμβάλλει τα μάλα στην Αμισόμ, ε, στην Αφρικανική Δύναμη στη Σομαλία ε, και επίσης είναι και επιφαλής της ΙΓΑΤ δηλαδή ε, των τοπικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπόλεμων μερών στο Νότιο Σουδάν. Προωθούμε τον πολιτικό διάλογο στην Αιθιοπία κυρίως αναφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα πιο εξειδικευμένα θέματα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε ενισχυθεί αυτή η εταιρική σχέση μέσα από διάφορες μορφές ε, διαλόγου ε, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αμυντόρων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι θέματα που έρχονται και επανέρχονται στις συζητήσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά την άποψή μας λοιπόν αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί ζωντανή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερσιά έχει το λόγο. για το Μαρόκο και την επιδείνωση της κατάστασης της καταστολής των δικαιωμάτων όσων είναι υπέρ των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοιτάξτε, μετά από τις απαντήσεις ε, για την ε, Αιθιοπία και με δεδομένη την κατάσταση στην Αιθιοπία και δεδομένη την κατάσταση στο Μαρόκο, αναρωτιέμαι τι απάντηση μπορείτε να μου δώσετε για το Μαρόκο γιατί η Αιθιοπία θεωρείται φυσιολογική χώρα, υποτίθεται, και με την οποία έχουμε υποτίθεται φυσιολογικές σχέσεις, ενώ είναι μία από τις χειρότερες δικτατορίες της Αφρικής. Ε, η απάντησή σας είναι απολύτως αναξιοπρεπής για την Αιθιοπία. Ζητώ συγγνώμη που δεν χρησιμοποιώ τη συνήθη διπλωματική γλώσσα, αλλά αυτό είναι το στυλ μου και ζητώ συγγνώμη που ασχολούμαι και που φυτρώνω εκεί που δεν με σπέρνουν για την Αιθιοπία, αλλά δεν αντέχω, πρέπει να το πω. Έρχομαι τώρα στο Μαρόκο. Έχουμε λοιπόν λοιπόν τα, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεγάλες μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις έχουν εκφράσει επανειλημμένως τις ανησυχίες τους για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση και κυρίως οι ΜΚΟ που ασχολούνται με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Μαροκινή, ο Μαροκινός Σύλλογος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά και το σκέλος το Μαροκινό της Διεθνούς Αμνηστίας συχνά αναφέρονται στις δωρεές, στην, ε, στην κατάσταση μη ισότητας, αποσύρουν τις δωρεές πολύ συχνά, ε, τη τελευταία στιγμή δεν τις κάνουν δεκτές η Καντίσα Ντεϊνή που πήρε το βραβείο των ΗΠΑ το 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μέρος από, είναι μία από τις προσωπικότητες τις συμβολικές που δείχνουν πόσο έχουν καταστρατηγηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μαρόκο. Ο Ζεν Μονμανί είναι νέος μποξέρ, θύμα βασανιστήριων θύμα επίσης των ε, διπλωματικών σχέσεων Γαλλίας και Μαρόκου. Είναι σύμβολο πολιτικού κρατουμένου. Θα μπορούσα να μιλήσω και για νέους φοιτητέ. Θα μπορούσα να μιλήσω για τους ακτιβιστές του κινήματος της 20 Φεβρουαρίου. Ε, πολύ μεγάλος κατάλογος, εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις μαροκινές φυλακές. Έχουμε ήδη αναφερθεί στο ζήτημα αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένε οι ερωτήσεις όλων μας και θέλω να μας απαντήσετε συγκεκριμένα και να μην μα πείτε τις συνήθεις λέξεις που μας λέτε, τις γενικέ. Έχουμε λοιπόν τη διαπραγμάτευση, τη διμερή ε, για την εταιρική σχέση με το Μαρόκο. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στον πυρήνα όλου αυτού του μηχανισμού και υπάρχει η βούληση να εμπλακεί η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Συγκεκριμένα παρακαλώ πείτε μου λοιπόν τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς στη διαπραγμάτευση αυτή θα ασχοληθείτε με τη δημοκρατία, με το κράτος δικαίου, με τη χρηστή διακυβέρνηση. Πώς. Και το αναφέρω ρητός, θα επιβεβαιώσουμε το ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Υποτίθεται, έτσι λέει το κείμενο, αλλά τελικά παρεποδίζονται οι ΜΚΟ να λειτουργήσουν, οι επικεφαλείς τους διώκονται, και καταστέλλονται κάθε φορά που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Ε, δεν γίνεται έτσι η δημοκρατία και δεν είναι αυτός ο ρόλος της οργανωμένης ε, κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις από πλευρά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Μπερνάχ ε, Σάβετς θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν είστε Άγγλος ή Γάλλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να πούμε ότι με το Μαρόκο διατηρούμε ένα διάλογο ανοιχτό, ειλικρινή και επικοδομητικό σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μαρόκο και μέσω του πολιτικού διαλόγου υψηλού επίπεδου. Πρόσφατα είχαμε την επίσκεψη του Επίτροπου Χάν το Δεκέμβριο του 2014 στο Συμβούλιο Σύνδεσης και μέσω το, της Επιτροπής Σύνδεσης και των διαφόρων υποεπιτροπών. Κυρίως τους ειδικού διαλόγους για, τον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται ενισχυμένος, στιβρημένος πολιτικός διάλογος και ο πολιτικός διάλογος γίνεται από τους διάφορους, ε, ε, διάφορα διευθυντικά στελέχη μας ε, θέλουμε λοιπόν να κάνει μεταρρύθμιση στον φάση επιχειρήσεις και να ε, κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από το νέο σύνταγμα του 2011. Αυτός ο διάλογος μακροπρόθεσμα θέλει να, ε, να διατηρήσει αυτές τις, αυτό το διάλογο που θα πρέπει να είναι ειλικρινής και επικοδομητικός και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, για ανθρώπινα δικαιώματα θα μεταβεί 28 και 29 Ιανουαρίου στο Μαρόκο και θα γίνουν συναντήσει με του διάφορου σημαντικού συνομιλητέ, ούτω ώστε να ακουστούν απόψει, να γίνει διάλογο στα ανθρώπινα δικαιώματα και να ανταλλαχθούν απόψει μεταξύ του, να εκφράσουμε τι θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκφράσουμε και τι ανησυχίε μα. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της 8ης συνεδριάσεως της Υποεπιτροπής ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα διακυβέρνηση που έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 2014 στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ερωτήματα και, και ζητήματα όσον αφορά τον περιορισμό των δραστηριοτήτων κάποιων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση ε, της κοινή των πολιτών στο Μαρόκο. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις είμαστε σε επαφή τακτική με το Εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχουμε και διάλογο τακτικό με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θέλουμε να ακούσουμε πώς αναλύουν αυτές την κατάσταση αλλά θέλουμε στο βαθμό του δυνατού να παράσχουμε στήριξη στις πρωτοβουλίες που εφαρμόζουν για να προωθήσουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα Όσον αφορά την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, η συνεργασία μας περνά κυρίως ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η, χρηματο... η χρηματοδότηση αυτού ε, ξεκινά από το 2014 και θέλουμε να απτυχθούν διάφορες δράσεις ε, Ανάπτυξη και ελέγχου από πλευρά τη κοινωνία των πολιτών των διαφόρων δημοσίων πολιτικών που εφαρμόζονται για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μα με την ε, κυβέρνηση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προσέγγιση μα είναι διαφανή, ενταξιακή και προβλέπει στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, κυρίως στα θέματα τη ισότητα και δίνουμε και οικονομική υποστήριξη όσον αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών και έχουμε ένα πρόγραμμα 45 εκατομμυρίων ευρώ πάνω σε αυτό με στόχο την υποστήριξη του σχεδίου της κυβερνήσεως για την ισότητα που εφέτηθηκε τον Ιούνιο του 2013. Στηρίζουμε επίσης τη χώρα σε θέματα δικαιοσύνης και οικονομικά. Στηρίζουμε τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα 70 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε ε, τη, τη, τη, τη Εθνικής για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, κάτι που εφετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και τα θέματα μετανάστευσης. Ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των μεταναστών. ύψος που διαθέτεται σε αυτό είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος 2014 υπεγράφει σχετική απόφαση. Να υπογραμμίσω και την θεσμική υποστήριξη που παρέχεται στη Βουλή των Εκπροσώπων του Μαροκινού Κοινοβουλίου. Εκεί δίνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε προγράμματα λοιπόν στήριξης και στηρίζουμε και το αντισιακό σχέδιο της Βουλής των Εκπροσώπων ε, κάτι που εγκρίθηκε τις αρχές του 2014. Επίσης, για 3 εκατομμύρια ευρώ, σε ένα ποστό 3 εκατομμύρια ευρώ, ανέρχεται η στήριξη τη Αθνοσυνέλευση του Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Διεθνού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Διπουργικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στα πλαίσια λοιπόν τη συνεργασία με το Μαρόκο, έχουμε ένα μέσο που πρέπει να υπογραμμιστεί στηρίζουμε και αυτή την μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Η επιτροπή αυτή παρέχει πολλές δυνατότητες για διπλωματικές ενέργειες, για ανταλλαγή απόψεων και διαλόγους ε, μεταξύ των εκπροσώπων των μοριτών των δύο χωρών. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος, τίθενται τα ζητήματα που εφήγησαν από το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου και πάντα θέτουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συνομιλούμε με τις αρχές του Μαρόκου στους διαφόρους διαλόγους που έχουμε στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών στο Μαρόκο κυρίως για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας μεγάλη είναι η στήριξη που παρέχουμε και μακράς διαρκείας και μέσω της ε, εφαρμογής του νέου συντάγματος του 2011 στηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται μέσω στεναρής υποστηρίξεως αυτών και μέσω χρηματοδοτήσεως των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών του Μαρόκου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Την οποία θα υποβάλω εγώ. Έχει να κάνει με το Καζακστάν. Γνωρίζετε ότι στις 27 Δεκεμβρίου, κατόπιν ετήματος της Ιντερπόλ, ο πολίτης Μουρατέκ και Τεμπαγεύ συνελήφθη στην Ισπανία. Είναι ένας από τους ε, επικεφαλείς της αντιπολίτευσης στο Καζακστάν. Ήταν στη Μαδρίτη γιατί ενδιαφερόταν για την κατάσταση άλλου αντιφρονούντος ε, από το Καζακστάν που ζητούσε πολιτικό άσυλο στην Ισπανία. Μιλούμε λοιπόν για δύο ανθρώπους που είναι επικεφαλής αν θέλετε της ε, αντιπολίτευσης ε, στο Καζακστάν. Ο κύριος Καζα... Και είχε έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας είχε μιλήσει για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Το ένταλμα βάσει του οποίου συνελήφθη ήταν διεθνές ένταλμα από την Ιντερπόλ. Το σκάνδαλο είναι ότι ο κύριος Κετεμπάγεφ έχει καθεστώς ασύλου. Ε, του έχει δοθεί άσυλο ε, στην Πολωνία και είναι πρωτοφανές αυτό. Κάποιος ο οποίος ε, έχει, του έχει δοθεί άσυλο σε μία χώρα να μπορεί να συλληφθεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελευθερώθηκε με την καταβολή εγγύησης, αφέθηκε ελεύθερος και το μόνο που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής είναι ακριβώς αυτό να αφαιθεί ελεύθερος από τις ισπανικές δικαστικές αρχές με την καταβολή εγγύησης. Δεν γνωρίζουμε όμως ποιες είναι οι δράσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θέλουμε να θέσουμε επιτάπητο σε αυτό το πρόβλημα και να ακούσουμε την άποψή σας, να μας πείτε λίγα λόγια για το τι κάνετε ήδη ή τι μπορείτε να κάνετε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει ο Άντρον και να είναι εδώ. Thank you, Madam Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν την ε, περίπτωση του κυρίου ε, Μουρατμπέκ και Τεμπάγεφ. Ο κύριος Κετεμπάγεφ, εξ όσων γνωρίζουμε, αφέθηκε ελεύθερο στις 15 Ιανουαρίου, αλλά εξακολουθεί να περιμένει μία δίκη για το κατά πόσον θα εκδοθεί ή όχι. Υπάρχει μια διμερή συμφωνία περί εκδόσεως ε, ανάμεσα ε, σε κράτος μέλους και μια τρίτη χώρα. Η δική μας υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και θέλω να σας πω ότι η υπηρεσία μας ε, παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Έχουμε καλέσει το Καζακστάν να σέβεται τις διεθνείς του υποχρώσεις. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεμονωμένων περιπτώσεων εξετάζονται σε πολλά επίπεδο και στο πλαίσιο του διαλόγου που υπάρχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται, τελειώνει ο χρόνος των ερωτήσεων. Έχουμε στη συνέχεια συνάντηση διευρυμένου Προεδρίου και εκεί θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμως να εκφράσω την προσωπική μου άποψη και απευθύναμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και σε εσάς και σε εσάς. Verán, eh, hemos, hemos establecido este, este tiempo de preguntas. Έχουμε προβλέψει λοιπόν αυτό το χρόνο ερωτήσεων έτσι ώστε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία όταν υποβάλλουν μια ερώτηση γνωρίζουν πολύ καλά την κατάσταση της χώρας για την οποία ε, υποβάλλουν ερώτηση. Η κυρία Βερσέα, για παράδειγμα, γνωρίζει άριστα τι γίνεται στο Μαρόκο, η κυρία Λοκμπίλερ γνωρίζει άριστα τι γίνεται στο Νεπάλ, ο κύριος Ντέμεσμέκερ γνωρίζει άριστα το τι γίνεται στην Ιγυρία. Επομένως, όταν, όταν ρωτούν οι βουλευτές, θέλουν πληροφορίες, ε, έτσι κάπως περισσότερες, ξέρουν τι γίνεται. Θέλουν κάτι πιο ουσιαστικό σαν απάντηση. Και σας λέω ότι κάνουμε αυτή την άσκηση εδώ πέρα και προσπαθούμε να μην ξεπερνούμε τα δύο λεπτά έτσι ώστε να είναι χρήσιμη αυτή η περίοδος ερωταποκρίσεων για τους βουλευτές. Δεν θέλουμε να μάθουμε ε, πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών, αλλά τι θα γίνει με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες αναφέρουν οι βουλευτές. Νομίζω ότι θα βελτιωθεί το επίπεδο της συνεδρίας αυτής των ερωταποκρίσεων. Θα καταλάβετε περισσότερο τι ζητούμε. Ε, για εμάς είναι κάτι το απαραίτητο και άλλωστε όλοι συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ε, τα λέω αυτά για να τα έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ. Περνούμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα μιλήσουμε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 Σήμερα το απόγευμα, δεν ξέρω τώρα από πού προέρχεται αυτός ο θόρυβος, λέει η Πρόεδρος. Α, προσπαθούμε να αποκτήσουμε σύνδεση με τη Βηρητό. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Άντεμς. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα άτομα χωρίς ηθαγένεια, αν ηθαγενείς. Είναι μία από τις ε, περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το ποιες είναι οι συνθήκες τις οποίες ε, ε αντιμετωπίζουν 60.000 από αυτούς είναι στην Ευρώπη, απάτριδες ή ανιθαγενείς. Καλό είναι να ακούσουμε πρώτα τη μελέτη και στη συνέχεια την εμπειρογνώμονα στη Βηρετό, αλλά δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη σύνδεση μέχρι τότε, να, να ακούσουμε πρώτα ε, τη Βηρετό, να κάνουμε πρώτα τη σύνδεση. Έχουμε χρόνο, ωραία. Θα παρουσιάσουμε πρώτα ε, την μελέτη της κυρίας Λάουρα Βανπάς από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στη συνέχεια θα συνδεθούμε ε, με τη Βηρητό. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνετε να παρουσιάσω τη μελέτη. Ελπίζω να είχα δυνατότητα να ζήξετε μια ματιά πριν έρθετε εδώ. Να σας πω ποια είναι η εμπειρία μας. Η εμπειρία μου από τη δεσκαλία που έκανα στο Πανεπιστήμιο Τόμπερ στην Ολλανδία ε, μιλώ για την ε, ιδεθαγένεια, και λοιπά τέτοια θέματα σε ε, φοιτητέ. Για πολλούς από αυτούς είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διάφορα συναφή προβλήματα και θεωρώ ότι αυτή το θέμα, το πρόβλημα της ανιθαγένειας τους βοηθά να μιλήσει κανείς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για κάποιον ανιθαγένεια θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία αναφέρεσαι και όταν μιλάς για αυτό αφορά βασικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είναι κάτι που είπαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθολική αξία και είναι κάτι που συγχωρίζει εμάς σαν ανθρώπινα όντα από άλλη κατάσταση και άλλα καθεστώτα. Και αυτό δοκιμάζεται σαν αξία όταν βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν ηθαγένεια, δεν έχουν υπηκότητα και δεν απολαμβάνουν τις προστασίες που απορρέει από μια συγκεκριμένη υπηκότητα. Ακόμα πιο σημαντικό, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με τους φοιτητές μου διερευνούμε ε, ένα ευρύ φάσμα άλλων προβλημάτων που άπτονται ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το φακό του απάτηδος. Λοιπόν, τι είναι να είναι κανείς ε, να έχει αυτό το πρόβλημα. Είναι ανθρώπινο, πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αυτός που δεν έχει ηθαγένεια δεν θεωρείται υπήκος κάποιου κατ' μέλους και δεν διαπέται από κανένα δίκαιο. Δηλαδή είναι κάποιος που δεν έχει υπηκότητα. Το δικαίωμα σε επικότητα είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Αν συζητούμε την κατάσταση που αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηθαγένεια, και και εκατοντάδες χιλιάδες στην Ευρώπη, αυτοί είναι άνθρωποι των οποίων τα δικαιώματα για επικότητα δεν ε, ικανοποιούνται. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό που συζητούμε. Αλλά πάει πολύ πιο βαθιά ο, ο συσχετισμός. Όταν βλέπουμε το θέμα αυτό της ανηθαγένειας είναι προϊόν πολλών άλλων προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γνωρίζουμε ίσως πολύ καλύτερα. Να δώσω κανένα δύο παραδείγματα από αυτό. Ε, Παραδείγματο χάρη, διάκριση κατά θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων μπορεί να εκδηλωθεί ποικιλοτρόπως περιθωριοποίηση, αποκλεισμό, ε, στιγματισμό. Ε, επίσης μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση, η στέρηση της υπηκότητας και να συμβάλλει στο να γίνει κανείς άπατρης. Δηλαδή διάκριση κατά των γυναικών ε, μπορεί να επηρεάσει το θέμα αυτό της ανηθαγένειας. Έχουμε πάρα πολλές χώρε όπου δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα οι γυναίκες να περάσουν υπηκότητα στα παιδιά τους όπως οι άντρες. Αν ο πατέρας είναι άγνωστος, δεν έχει ηθαγένεια, δεν μπορεί να περάσει την ηθαγένεια ε, δημιουργείται θέμα στο δίκαιο ανισότητα των φίλων, όσον αφορά την θα και είναι κάτι που ε, διαιωνίζει το πρόβλημα αυτό. Με τους φοιτητέ μου εξετάζουμε πώς η ανηθιαγένεια είναι και αίτιο και καταλήτης για πολλά άλλα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι προβλήματα τα οποία ίσως γνωρίζουμε πολύ καλύτερα. Η εθνικότητα, ξέρουμε, ανοίγει την πόρτα σε πολιτική συμμετοχή. Ε, για μια δημοκρατία, για να είναι ενταξιακή δημοκρατία, για να έχει νόημα για όλους σε μια κοινότητα, σε μια κοινωνία, πρέπει να έχει κάνει το δικαίωμα να συμμετέχει. Αν κανείς δεν έχει ηθαγένεια, έχει πρόβλημα. Στην πράξη λοιπόν η υπηκοότητα ανοίγει και την πόρτα στο να απολαμβάνει κανείς πολλά άλλα δικαιώματα. Αν δούμε ποια είναι η κατάσταση των παιδιά που δεν έχουν ηθαγένεια, έχουν πρόβλημα να γραφούν στα μητρώα γεννήσεων, ε, περίθαλψη, να τελειώσουν το σχολείο. Αν δούμε τι γίνεται με του ενήλικε που έχουν το ίδιο πρόβλημα, δεν μπορούν να μπουν επίσημη, στην επίσημη αγορά εργασία, να ανοίξουν λογαριασμό στην τράπεζα, να έχουν ιδιοκτησία, να κληρονομούν ιδιοκτησία, να έχουν κοινωνική ασφάλιση, να παντρευτούν, να ταξιδέψουν. Οπότε αυτή η ανηθαγένεια δημιουργεί πολλά άλλα προβλήματα τα οποία μας ε, προβληματίζουν, μας και τα Μπορεί να οδηγήσει σε καταναγκαστικό εκτοπισμό, σε κράτηση, μπορεί κανείς να είναι ευάλωτος σε εκμετάλλευση και μπορεί να είναι και αντικείμενο εμπορίου. Έχει γίνει μια μελέτη. Μελέτη μάλλον θα ξεκινήσει το επόμενο μήνα. Την ανέλαβα εγώ με κάποιου συναδέλφου που εξετάζει συγκεκριμένα τη διασύνδεση μεταξύ ανιθαγένειας και εμπορίου ανθρώπων. Μελετά τι γίνεται με του ηθαγενείς, με του ντόπιου στην Ταϊλάνδια που εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανιθαγένειας δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος εμπορίου ανθρώπων ε, διότι υπάρχουν ε, περισσότερα αίτια ε, για να γίνει αυτό το εμπόριο ανάμεσα στους απάτηδες. Είναι πιο φτωχοί αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν καλή εκπαίδευση εν συγκρίση με τους γείτονες που έχουν την ηθαγένεια. Δεν έχουν πρόσβαση στις δομές για στήριξη κρατική. Αν τελικά είναι αντικείμενα εκμετάλλευση, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις κρίσεις, να τις αντιμετωπίσουν τις προσωπικές και τις οικονομικές και μπορεί τελικά να βρεθούν σε θέση εκμετάλλευση πιο γρήγορα από τους άλλους. Βασικά λοιπόν, μετά από 12 εβδομάδες μαθημάτων ε, με τους φοιτητέ μου, περίπου το Μάιο κάθε χρόνο, δεν μιλάμε μόνο για την Αθαγένεια, συζητήσαμε και τα θέματα των μειονοτήτων, των δικαιώματων των γυναικών, διακρίσεις, κράτος δικαίου, δικαιώματα παιδιών, μετανάστευση, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά δικαιώματα, υποχρεωτικός αυτοκτονισμός, εκδημοκρατισμός, συγκρούσεις, δημιουργία κρατών, πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, ο λόγος που σας τα λέω όλα αυτά ποιο είναι Βλέπετε η έκθεση που σας παρουσιάζω ανοίγει με παρόμοια εισαγωγή. Γιατί, Γιατί είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε συζήτηση για δράση αντιμετωπίσεως του προβλήματος στο σωστό πλαίσιο. Ε, πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, διαφορετικά προβλήματα, χρειάζονται την προσοχή μας και η αδίποτε πρόοδος μπορεί να είναι δύσκολη. Σε αυτό το περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα θέμα όπως είναι η νηθαγένεια ε, που δεν ήταν πολύ ορατό και δεν έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από την ε, διεθνή κοινότητα τελικά να γίνει κάτι ελκυστικό και να το προσέξουν. Αλλά δεν θα πρέπει να εκλειφθεί σαν κάτι που είναι καινούριο ή συμπληρωματικό Επί μακρόν υπήρχε σαν πρόβλημα, επηρεάζει και πολλέ άλλε προτεραιότητε σχετικέ με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε η καταπολέμηση της ανιθαγένειας είναι και καταπολέμηση άλλων προβλημάτων ανθρωπινών δικαιωμάτων είναι μια μάχη στην οποία ήδη έχουμε επιδοθεί. Παραδείγματο χάρη να προωθήσουμε ισότητα των φύλων σε όλου του τομεί του νόμου, τη νομοθεσία, θα βοηθήσει να προωθηθεί η αποφυγή του φαινομένου τη ανηθαγένεια. Έτσι, δεν περαιτέρω η καταπολέμηση άλλων προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί επίση να στηριχθεί εάν αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά δικαιώματα, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι υποβόσκετες παράγοντες που ε, ε, μπορεί να συμβάλλουν στον αποκλεισμό. Τούτων λεχθέντων η ανηθαγένεια δεν είναι κάτι καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε θα πρέπει να ειδωθεί σαν κάτι ξεχωριστό από άλλα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπω δείχνει και η έκθεση, εκεί εντοπίζεται σελίδε 18 μέχρι 19 ότι υπάρχουν διάφορε ξεχωριστέ διασυνέσει μια και προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προανέφερα τι συνέσει μεταξύ ανηθιαγέννη, ισότητε των φύλων, προστασία των μειονοτήτων, θρησκευτικέ ελευθερίε, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά δικαιώματα και εμπόρια ανθρώπων αλλά είναι η ηθαγένεια επίση. Είναι και μια πρόκληση και πρόβλημα σχετίζεται με την πρόσφαση των δικαιωμάτων των παιδιών, με τη δημοκρατία και με το έργο των προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι χρειαζόμαστε, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των διασυνδέσεων και προσεκτική αναθεώρηση του τι άλλε προσπάθειε γίνονται και να δούμε τι μπορούμε να στηρίξουμε, πού μπορούμε να το επεκτείνουμε. Ε, πρέπει να καταλάβουμε τι ήδη έχει γίνει. Πρέπει να βρούμε τομείς στους οποίους είναι δυνατόν να αυξήσουμε διμερή ή πολυμερή προσπάθεια. Τι θεσμικές ρυθμίσεις απαιτούνται για να επιτευχθεί αυτό. Βασικά, περί αυτού πρόκειται η έκθεση. Κάνει μια επισκόπηση υφισταμένων προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα πλαίσια της δράσης, της εξωτερικής δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να συναγάγει συμπεράσματα για να προχωρήσουμε. Θέλω ακροθυγώς να αναφερθώ σε πέντε χαρακτηριστικά της εκθέσεως που ελπίζω ότι θα διαρευνήσετε περαιτέρω μετά την συνεδρίαση. Ε, λοιπόν, καταρχάς η έκθεση εξετάζει το ζήτημα της ανηθαγένειας από την έποψη της εσωτερικής διαστάσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εστιάζεται βασικά επί εξωτερικής δράσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δοθήσεις όμως τη σημασία συνοχής μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσεως για τα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η έκθεση φωτογραφίζει και το θέμα της ανιθαγένειας εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βλέπουμε ότι πράγματι δύο χώρες από τις δέκα μεγαλύτερες έχει τις είναι ε, τα δύο χώρε που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την ηθαγένεια είναι χώρε Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Υπάρχουν άλλε χώρε όπου έχουμε χιλιάδε άτομα με αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει σημαντικό πληθυσμό ανθρώπων εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω με αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε επίση ότι υπάρχουν σοβαρέ συνέπειε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε άλλη έκθεση. Δημοσιεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εθαγένεια. Ακόμα χωρίς ηθαγένεια, ακόμα υποφέρει είναι ο τίτλο και δείχνει διάφορα είδη προβλημάτων ανθρώπινα, προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εντοπίζουν αυτοί οι άνθρωποι εντό τη Ευρώπη και εντό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Προβλήματα παρατεταμένης κρατήσεω, ε, μεγάλης φτώχειας ε, και ανθρώπων που έχουν ε, πέσει σε ένα νομικό κενό. Άρα η ανηθαγένεια είναι και θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υλοποίηση των προσδοκιών των περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με αυτά υπόψη η έκθεση αναφέρεται σε κάποιες σημαντικές εξελίξεις εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως δεσμεύσεις όσον αφορά καθολική πρόσβαση στη σύμβαση του ΟΗΕ για τους απάτηδε και τα συμφέροντα και το συντονισμό των κρατών μελών για την προστασία τους όσον αφορά τα άτομα με, που έχουν το πρόβλημα της ανηθαγένειας σχετικά με τη μετανάστευση. Μέχρι τώρα ήταν κατά περίπτωση αντιδράσει. Χρειάζεται πιο συνεκτική, ε, συντονισμένη αντίδραση για το πρόβλημα αυτό της Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Και αυτό με τη σειρά του θα είναι κάτι σημαντικό για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία για, για αυξημένη εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Βλέποντας την εξωτερική δράση τώρα, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η ανηθαγένεια δεν αποτελεί συγκεκριμένη προτεραιότητα προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλα αυτά, η ανηθαγένεια εντοπίζεται σαν ένα τομέα ιδιαίτερη ανησυχία σε κάποια στατηγικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και τη σφαιρική προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την κινητικότητα και τη μετανάστευση. Λοιπόν, ποια είναι η πρόκληση, να εντοπίσουμε τρόπου με του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει προσπάθειε αντιμετώπιση του προβλήματο ανηθαγένεια, διότι συχνά και σε αυτά τα θέματα κρύβονται. Γιατί το λέω αυτό, δηλαδή η προσπάθεια σχετίζεται με συναφή προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι με αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, το συγκεκριμένο. Βλέπουμε προγράμματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ισότητα των φύλων σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου και του νόμου για την υπηκότητα. Υπάρχουν καταστάσεις κατά τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκεί ε, αναφέρονται τα προβλήματα της ανιθαγένειας. Αν δείτε όλες αυτές τις προσπάθειες μέχρι τώρα, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει, χρειάζεται να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να προωθηθεί το όλο θέμα Υπάρχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Υπάρχει προσπάθεια να αυξηθεί η προστασία όσον αφορά τα άτομα ε, που έχουν προβλήματα ελλείψης ανιθαγένειας, να μειωθούν οι περιπτώσεις ανιθαγένειας και όπου έχει καταβάλει προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι στον κόμβο διασύνδεσης με άλλα θέματα που αποτελούν προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, δικαιώματα παιδιών, ισότητα των φίλων, ε, ανεξιθρησκεία. Λοιπόν, η έκθεση συνεχίζει και κάνει κάποιες συστάσεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να ισχύσουμε πολυμερή και διμερή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το θέμα της ανιθαγένειας. Θέλω λοιπόν να τονίσω ένα δω πλαίσιο της σελίδας 29 της εκθέσεως. Εκεί βλέπετε κάποιες ιδέες. Αυτές αφορούν τι δυνατότητε και ευκαιρίε που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει προσπάθεια καταπολέμηση του φαινομένου τη ανηθαγένεια. Βλέπουμε λοιπόν πολλά θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί το Κοινοβούλιο έχει θετήσει θεματικά ψηφίσματα, έχει για ακροάσει, έχει κάνει επισκέψει σε κάποιες χώρε να δει ποια είναι η κατάσταση αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτόπου ή ε, συνεργάζεται με άλλου βουλευτές σε όλο τον κόσμο, ούτω ώστε να βρεθεί ε, να ισχυροποιηθεί αντίδραση άλλων κοινοβουλίων στον αφορά τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε σε συγκεκριμένο θέμα τη ανηθαγένεια. Συνεχίζει η έκθεση. Αναφέρει θεσμικέ διευθετήσει που θα μπορούσαν να στηριχθούν και να ενισχυθούν. Παραδείγματο χάρη, αναφέρονται εργαλεία, κατάρτιση, δυνατότητε υποβολή καταγγελιών που χρειάζεται ενίσχυση όλα αυτά. Και αναφέρεται και με ενδεχόμενη βάση, ούτω ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί ένα τέτοιο εργαλείο ε, και να μπορεί τάχιστα να εντοπίζει τα προβλήματα σε διάφορες χώρες. Να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να καταβάλει προσπάθειες όσον αφορά να διεξαγάγει διάλογο με συγκεκριμένες χώρες που υπάρχουν τα προβλήματα και να αντιμετωπιστεί το θέμα της ανηθαγένειας σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Η έκθεση τελικά κλείνει στις τελευταίες σελίδες αναφέροντας κάποιες προτεραιότητες θεματικές και κατά χώρα. Εκεί αναφέρονται τα μαθήματα που έχουμε συναγάγει για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτά τα μαθήματα τα εφαρμόσαμε σε εξελίξει στον τομέα της ε, ανηθαγένεια. Ο Μάρκ Μάλι από την ΥΠΑ Τερμοστία του ΟΗΕ θα ακούσει κάποιε συγκεκριμένε δυνατότητε που παρουσιάζονται. Είναι η εκστρατεία τη ΥΠΑ της του ΟΗΕ για να θεθεί τέρμα στο πρόβλημα. Αναφέρεται η έκθεση και στη διεθνή εκστρατεία να θεθεί τέρμα στην ε, διάκριση των φύλων στι νομοθεσίε για καθώς και κάποιες χώρες όπου τώρα υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες να γίνει διαφορά όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος ενηθαγένειας και χώρες όπου η ενηθαγένεια αρχίζει να αναδύεται σαν ένα καταπήγον θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν ερωτήσεις για δίποτε από αυτά, ε, με τα χαράς να απαντήσω. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ομάιλη, επικεφαλής του Τμήματος για την Ανηθαγένεια στην Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκτός από την εντολή που έχουμε να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες, έχουμε και εντολή να προστατεύσουμε τους ανιθαγενείς. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ σήμερα. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων είναι κάτι το σημαντικό για εμάς, διότι οι βουλευτές σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου ε, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, γιατί πολύ συχνά το πρόβλημα έχει να κάνει με την νομοθεσία, με την ψήφιση αυτής, με την ύπαρξη αυτής ή την εφαρμογή αυτής. Νομίζω ότι έχετε γραπτό αντίτυπο ε, στα αγγλικά της παρουσίασης PowerPoint που ε, έχω και μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Στις 4 Νοεμβρίου του 2014 ο Αντώνιο είπε τους αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία έτσι ώστε να μην υπάρξει πλέον ανιθαγενής άνθρωπος μέσα σε 10 χρόνια. Είναι πολύ φιλόδοξος αυτός ο στόχος. Πιστεύουμε όμως ότι αν αποτελέσει στόχο ε, της διεθνούς κοινότητας οι ηγέτιδες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών, η παγκόσμια κοινότητα στο σύνολό του θα αρχίσουν να συνεννοούνται περισσότερο για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό. Και είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μας αφορά όλους σήμερα και θα ήθελα να σας υπογραμμίσω ορισμένα γεγονότα. Πρώτον, η Πάρα πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται από αυτό. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι ανιθαγενείς και εκτός από τους ανιθαγενείς, ορισμένοι ανιθαγενείς αναγκάστηκαν ε, εκτός από το ότι είναι ανιθαγενείς, τους ανάγκασαν να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν προστασία ως πρόσφυγες στο εξωτερικό. Το άλλο θέμα είναι ότι πολλές τέτοιες καταστάσεις έχουν χρονίσει, έχουν παραχρονίσει. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, γνωρίζουμε ότι Υπάρχουν 600.000 ανιθαγενείς άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί από αυτούς είναι ανιθαγενείς για περισσότερα από 20 χρόνια και σίγουρα αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, γνωρίζουμε ότι η διάκριση είναι σημαντικό πρόβλημα και πολύ συχνά η αιτία. Η διάκριση εναντίον των γυναικών των ε, μειονοτικών πληθυσμών ενώ πολύ συχνά ε, βλέπουμε ότι ε, εμπεριέχονται εκεί ζητήματα φυλής ή εθνότητας. Και πολύ σημαντικό είναι ο στα παιδιά. Έχουμε εκτιμήσει ότι γεννιέται ανιθαγενές παιδί, ένα ανιθαγενές παιδί γεννιέται, κάθε δέκα ε, λεπτά στις ε, πέντε πιο σημαντικές χώρες του κόσμου σε σχέση με το θέμα αυτό. Ποιες είναι, ποια είναι τα εμπόδια για τις λύσεις. Για να το εξηγήσω, να επιλύσουμε το πρόβλημα της ανηθαγένειας χρειάζεται κατά 80% πολιτική βούληση και μόνο κατά 20% ε, τεχνική δυνατότητα, τεχνογνωσία και πόροι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει παραγνωριστεί, έχει παραμεληθεί και πολύ συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει η ανισαγένεια. Εξού και ξεκινήσαμε αυτή την εκστρατεία στις 4 Νοεμβρίου του 2014. Στην αρχή ξεκινήσαμε με την έκδοση ειδική ε, έκθεσης η οποία εξηγεί το πρόβλημα τι είναι η ανηθαγένεια, πώς πλήττει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Ο Αντώνιο Γκουτιέρης, ο ύπατος αρμοστής, στη συνέχεια εξέδωσε μια δημόσια επιστολή την οποία υπέγραψαν ε, πάρα πολλές ε, προσωπικότητες από όλο τον κόσμο βραβευθέντες ε, με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης όπως ο Ντέσμον Τούτου μεταξύ άλλων όλοι οι συνυπογράφοντες καλούν τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και τρίτον, έχουμε εκδόσεις την είπατε αρμοστία. Έχουμε καταρτήσει μάλλον ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης το οποίο απαριθμεί τους τρόπους με τους οποίους τα κράτη μπορούν να, οι κυβερνήσεις μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα και ορισμένα από τα βήματα έχουν να κάνουν με την επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων ανηθαγένειας τα οποία ε, υπάρχουν εδώ και 10-20 χρόνια ενώ άλλα βήματα έχουν να κάνουν με την εξέταση των αιτιών για τις οποίες υπάρχει ανηθαγένεια και πώς μπορεί να υπάρχει πρόληψη αυτού του φαινομένου π.χ. διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί που γεννιέται σε μια χώρα και δεν μπορεί να έχει άλλη ηθαγένεια να έχει τουλάχιστον την ηθαγένεια της χώρας στην οποία γεννιέται και θα πρέπει να απαλείψουμε τις διακρίσεις με βάση την εθνότητα στο τομέα της ηθαγένειας ή της υπηκοότητας μπορεί να σας εκκλείσει αλλά παραμένει πρόβλημα σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο και γιατί πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να εξαλειφθεί το πρόβλημα αυτό μέσα σε μία δεκαετία. Θα σας μιλήσω για ορισμένες εξελίξεις οι οποίες μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Αν δούμε τι έγινε τα τελευταία 12 χρόνια, τότε καταλαβαίνουμε ότι ορισμένες κυβερνήσεις πράγματι έχουν αναλάβει δράση. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον Τέσσερα εκατομμύρια ανιθαγενείς έχουν αποκτήσει ηθαγένεια από το 2003 μέχρι σήμερα. Άρα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών και ελπίζουμε ότι και οι άλλες κυβερνήσεις θα δουν ε, την πρακτική και την εμπειρία των συγκεκριμένων χωρών και θα την υιοθετήσουν. Δεύτερον, πάρα πολλές χώρες έχουν μεταρρυθμίσει τον εθνικό τους νόμο περί ηθαγένειας και μάλιστα νόθηκε μια υπουργική διάσκεψη στη Γενέβη το 2011 στην οποία 12 περίπου χώρες είπαν ότι θα καταργήσουν νομοθεσία η οποία επιβάλλει διακρίσεις και έτσι μεταξύ άλλων θα αποφύγουν ε, το ενδεχόμενο παιδιά να μην έχουν ηθαγένεια. Είναι μια εξέλιξη αυτή λοιπόν. 12 χώρες έχουν μεταρρυθμίσει την εθνική νομοθεσία έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν το ίδιο νομικό δικαίωμα να μεταδώσουν την ηθαγένεια στο παιδί τους όπως και οι πατέρες οι μητέρες όπως λοιπόν και οι πατέρες. Υπάρχει μια τάση δηλαδή μεταρρυθμιστική ε, παντού στον κόσμο η οποία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική. Και τέλος να σας αναφέρω ότι, είναι, ότι υπάρχουν δύο βασικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν αυτό το θέμα, η σύμβαση του 61 και η σύμβαση του 54. Τις είχαμε ξεχάσει πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια όμως έχουν έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον στις συνθήκες αυτές. 45 χώρες προσχώρησαν ε, σε αυτές τις συνθήκες, τις κύρωσαν και τις αφομοίωσαν αν θέλετε και ε, τον επόμενο χρόνο, χρόνο και άλλες χώρες θα, τις, ε, θα προσχωρήσουν σε αυτές. Άρα υπάρχει δέσμευση να αναλυθεί δράση. Τώρα, χρειάζεται περισσότερη πολιτική βούληση, αυτό το είπα. Κάτι το εθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η ανιθαγένεια συνεχώς βρίσκεται στην διεθνή πολιτική ατζέντα. Το τελευταίο ε, ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη δράση της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες καλωσορίζει τη δράση της υπηρεσίας μας για την εξάλληψη του φαινομένου μέσα σε 10 χρόνια. Ε, αυτό συζητείται και... Αυτό συζητείται και στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τίθενται αυτές οι ερωτήσεις στο πλαίσιο της ε, περιοδικής αναθεώρησης της κατάστασης ε, παγκοσμίω. Επομένως, αυτά είναι όλα πολύ ενθαρρυντικά για να δούμε πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προσπάθεια. Θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εθετήσει ένα ψήφισμα για την ανιθαγένεια και να στηρίζει το κάλεσμα το δικό μας της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες έτσι ώστε να λήξει, να εξαλειφθεί το φαινόμενο μέσα σε 10 χρόνια και θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει ένα κράτος μέλος να ε, δείξει το δρόμο, ε, να δείξει το καλό παράδειγμα να καλέσει όλα τα κράτη-μέλη να δείξουν το καλό παράδειγμα έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν σε αυτές τις συμβάσεις, να προστατεύσουν τους ανηθαγενείς και να προλάβουν τέτοια φαινόμενα πριν από την εμφάνισή τους, αλλά και να επιλύσουν τα υφιστάμενα προβλήματα. Θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει, ε, να ζητήσει να εξεταστεί το θέμα της ανισαγένειας και το πώς αντιμετωπίζουν οι χώρες που έχουν αιτηθεί να προσχωρήσουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι έχουμε έναν απρόσκοπτο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Εξωτερική Δράση. Θα μπορούσε να κάνει διάφορα βήματα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υιοθετήσει ένα πλαίσιο έτσι ώστε η ανηθαγένεια να εξετάζεται στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το είπε άλλωστε θα το έκανε το 2012, και συστηματικά η ανιθαγένεια να περιλαμβάνεται στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να χρηματοδοτήσει δράσεις σε όλο τον κόσμο της, των ΜΚΟ, της υπατής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις στο θέμα αυτό και θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τέλος να συμπεριλάβει το πρόβλημα αυτό στους αναπτυξιακούς στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015. Αυτά είναι τα ζητήματα που επιθυμούμε να συζητήσουμε περισσότερο με εσάς. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε σύνδεση με τη διάσκεψη ο κύριος Ραντζή Πενσαλάμ, μέλος του προεδρίου ε, του Γραφείου μάλλον, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, των Παλαιστίνιων προσφύγων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να με ακούτε. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους σας, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλους τους ε, εμπειρογνώμονες των ε, κρατών μελών και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάποιες ε, απόψεις ε, δικές μου σχετικά με τη μελέτη της κυρίας Βάμπας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία προβάλλει πάρα πολλά θέματα που διακυβεύονται σχετικά με την ανιθαγένεια και την ε, καταγραφή εκγενετής. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα θέματα και στα προβλήματα που υπάρχουν. Ένα λοιπόν από τα ε, θέματα που έχει σχέση με τη νομοθεσία και τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας είναι ότι στον δικό μου τον τομέα ε, όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση των ε, Παλαιστινίων προσφύγων. Όσον αφορά την ανηθαγένεια στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε διάφορες χώρες και νομίζω ότι εσείς τα γνωρίζετε τα θέματα αυτά καλύτερα από εμένα. Επίσης, θα ήθελα να συζητήσουμε για το θέμα της ε, ανηθαγένειας ε, σχετικά με τους πρόσφυγες. Αν δούμε λιγάκι τη Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία, βλέπουμε πώς αντιμετωπίζεται η έννοια του πρόσφυγα. Και βλέπουμε επίσης πώς ε, περιπλέκεται η κατάσταση αλλά και η ζωή των Παλαιστινίων προσφύγων. Και όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Διότι η ανιθαγένεια δεν ξεκινάει με την καταγραφή εκγενετής. Κάποια στιγμή γίνεται μια καταγραφή, οι ε, περιπλοκές προκύπτουν από το νομικό καθεστώς και τις ε, προεκτάσεις τους. Ε, κυρίως στο Λίβανο αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι το θέμα των δικαιωμάτων. Η κατάσταση είναι τόσο τραγική μετά από 67 χρόνια εξακολουθούν πολλοί να είναι πρόσφυγες η κυβέρνηση του Λιβάνου μερικές φορές τους αντιμετωπίζει ως πρόσφυγες, ε, άλλες φορές πάλι ως αλλοδαπούς. Μας περιπτώσει αυτό σημαίνει υποβάθμιση των δικαιωμάτων τους και έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολλές ε, κοινοοικονομικές ε, φρικαλαιότητες, έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα. Τώρα στο Λίβανο οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες δεν έχουν ας πούμε το δικαίωμα ιδιοκτησίας, δεν έχουν ηθαγένεια προφανώς γιατί είναι πρόσφυγες Μία δυσκολία λοιπόν που προκύπτει από αυτό έχει σχέση με το δικαίωμα στην εργασία, τα κοινωνικά δικαιώματα, ας πούμε το δικαίωμα στην εργασία. Και εμείς ε, προσπαθούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις έτσι ώστε να ενταχθούν οι Παλαιστίνοι στις κοινωνίες και όχι να περιθωριοποιηθούν. Παρόλα όλα αυτά ε, σας λέω ότι το πρόβλημα λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις διότι το νομικό καθεστώς που απολάβουν είναι απαράδεκτο, είναι πρόσφυγες και το τι είναι ένας πρόσφυγας, ένας πρόσφυγας είναι ανιθαγενής και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Οι απελιστήνοι πρόσφυγες ε, δεν έχουν ε, πρόσβαση στην επανεγκατάσταση. Όποιος έχει γεννηθεί στην Ιορδανία, παραδείγματος χάρη ή στο Λίβανο, ε, πρέπει να καταγραφεί. Βέβαια οι ίδιοι είναι επιφυλακτικοί γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα έχουν καμία ελπίδα να επαναγκατασταθούν στην ε, πατρίδα τους. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων σε άλλες χώρες. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω της κρίσης στη Συρία. Όπως γνωρίζετε οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες που βρίσκονται στη Συρία και διαφεύγουν σε άλλες χώρες όπως την Ιορδανία και το Λίβανο εξακολουθούμε να βρίσκονται υπό την αιγίδα της Ούνρα, όμως υπάρχει λάθος ερμηνεία του άρθρου Δέλτα που ε, αποκλείει τους Παλαιστινίους από τις υπηρεσίες της Ούνρα γιατί αυτοί θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται από τις ε, διατάξεις ε, από το άρθρο D Πρέπει λοιπόν αυτό το άρθρο να επανεξεταστεί για να δούμε ε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που είναι τεράστιο. Η Ούνρα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να βοηθήσει σε περίπτωση αιτήματος ε, επαναγκατάστασης ε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η κρίση ως εκ τούτου θα πρέπει να λάβει η χώρα ουσιαστικός διάλογος για όλα αυτά τα θέματα και για το πώς μπορούμε να ανακουφίσουμε λιγάκι αυτούς τους πρόσφυγες που τώρα έχουν εγκαψαθεί στη Συρία ε, και προσπαθούν να φύγουν σε άλλες χώρες. Στην Κύπρο βρίσκονται πάρα πολλοί πρόσφυγες ε, και μιλάμε για περίπου 200 άτομα που βρίσκονται στην Κύπρο έχουν ε, εγκλωβιστεί εκεί και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όπως ας πούμε την επανένωση των οικογενειών και άλλα. Ε, όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι απάτριδες όταν ε, βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμούν να εγκαψαθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αυτά τα εμπόδια που δημιουργούν οι χώρες της ε, Ευρώπης και αυτά τα εμπόδια ε, δυσχεραίνουν περαιτέρω τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Επίσης ε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, κάποιες προτάσεις ε, δικές μου. Θα ήθελα λοιπόν να πω την εξής πρώτη μου πρόταση. Οι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα και μέσω της ε, υπηρεσίας εξωτερικής ε, δράσης είναι ευπρόσδεκτες αλλά κατ' ουσίαν η κατάσταση των παιδιών δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Ας πούμε, οι απάτριδες από τη Συρία, όπως και κάποιοι Κούρδοι και Παλαιστίνοι, αυτοί έχουν το μεγάλο πρόβλημα πρόσβαση σε διεθνή προστασία και όχι τόσο της ηθαγένειας. Γιατί σας λέω, το πρόβλημα δεν είναι κατ' ουσίαν η ηθαγένεια, αλλά η στέρηση δικαιωμάτων. Γιατί ακόμα και αν χορηγηθεί η ηθαγένεια, δεν αλλάζει τίποτα το σπουδαίο. Ε, υπάρχουν ε, προβλήματα που επηρεάζουν τα πάντα και όλους. Αυτό λοιπόν που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί είναι διεθνή προστασία. Το δεύτερο που χρειάζονται είναι τα κοινωνικά τους δικαιώματα, ανεξάρτητα από την ηθαγένεια. Ε, στη Συρία υπάρχουν οι Παλαιστίνοι, απάτριδες πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν σε με το Λίβανο κάποια πρόσβαση σε κάποια δικαιώματα ή είχαν στο παρελθόν τώρα όμως λόγω του πολέμου έχει επιδεινωθεί κατά πολύ η κατάστασή τους. Ε, μία δεύτερη σύσταση που θέλω να κάνω έχει σχέση με την πρόσβαση σε διεθνή ε, προστασία ε, πάντα μιλάμε για τους Παλαιστίνιους. Η UNHCR θα πρέπει να σέβεται την σύμβαση περί προσφύγων και θα πρέπει μάλιστα να την συμπεριλαμβάνει και στις ε, συστάσεις της. Αυτή τη στιγμή κανένα κράτος μέλος ε, δεν ερμηνεύει σωστά το άρθρο 1D που αφορά τους Παλαιστινίους οι οποίοι έχουν ε, καταθέσει έτσι για άσυλο και αυτοί που έχουν εκδοχθεί, εκδοχθεί από τη Γάζα. Συμπεριλαμβάνονται και αυτοί όπως προβλέπεται και στη σχετική σύμβαση του 51. Οι Παλαιστίνοι ως κοινότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο και επίσης ε, θα πρέπει να έχουν την ε, δυνατότητα οι απάτριδες, ε, κυρίως οι Παλαιστίνοι, να εγκατασταθούν, να απολαύουν αυτού του δικαιώματος. αν δεν υπήρχε η κατάσταση στη Συρία, η Παλαιστίνη δεν καλύπτονται από την ε, Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, το UNHCR. Πάντως αυτό θα πρέπει να είναι ειδικό θέμα που ε, οφείλουμε να το εξετάσουμε ιδιαίτερα σε σχέση με τους Παλαιστίνιους. Μία άλλη σύσταση που έχω να κάνω αφορά το θέμα της ε, ανιθαγένειας ε, σε σχέση με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διευκολύνται τουλάχιστον οι συζητήσεις ε, της UNHCR κυρίως σε σχέση με την UNRWA έτσι, έτσι ώστε οι Παλαιστίνοι από τη Συρία να έχουν δικαίωμα επαναγκατάστασης. Η κατάσταση στη Συρία είναι τραγική εκεί έχουν καταστραφεί ολόκληροι καταβλισμοί στη Συρία. Επίσης βλέπουμε ότι η κρίση πλέον έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που έχει οδηγήσει σε απόγνωση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μια άλλη σύστασή μου και παράδειγμα που δεν θέλω να φέρω είναι η κατάσταση των Παλαιστινίων από τη Συρία που έχουν ε, καταφύγει στην Κύπρο. Δεν έχουν ε, δικαίωμα προστασίας, βρίσκονται εν κενό κατά κάποιον τρόπο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, θα είχε αξία αυτή την έκθεση για την ανιθαγένεια να την προωθήσετε και σε σχέση με τους Συρίους που έχουν εγκλωβιστεί στην Κύπρο. Όπως γνωρίζετε η κατάσταση αυτή υπάρχει εδώ και πολλούς μήνες και είναι άμεσο αποτέλεσμα του ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι Παλαιστίνοι από τη Συρία δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαιώματα όπως σας είπα ούτε και το δικαίωμα της επαναγκατάστασης και δεν καταβάλλονται σχεδόν καθόλου προσπάθειες για επαναγκατάσταση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν με εκτιμήσεις περίπου 200 άτομα σε καταβλισμό. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι Παλαιστίνοι. Με συγχωρείτε διακόπτη πρόεδρος. Νομίζω ξέρετε θα πρέπει να ολοκληρώσετε σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Υπάρχει λοιπόν έλλειμμα ε, προστασίας των ε, ανιθαγενών και των οικογενειών τους και νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην επανασύνδεση των οικογενειών. Και με αυτή την κατακλίδα επιτρέψτε μου πράγματι να ολοκληρώσω την ε, παρέμβασή μου. Αν κάποιος έχει να υποβάλει κάποια ερώτηση, παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ παραμείνετε στη σύνδεση, μην κλείσετε σύνδεση. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ιωάννα Γκριν, Διευθύντρια της Οργάνωσης Εθνών και Λαών που δεν εκπροσωπούνται. Έχει έδρα εδώ στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μας κάλεσε εδώ να συμμετάσχουμε στην ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την ανηθαγένεια και τις συνέπειες που έχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για σας που δεν γνωρίζετε τη δουλειά μας, είμαστε διεθνής δημοκρατική οργάνωση, μια βία οργάνωση ε, και θέλουμε, προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνουμε μια πλατφόρμα για τους ηθαγενείς, τις μειονοτικές, ε, ε, μειονότητες και τους κατοίκους κατεχομένων περιοχών. Θα ήθελα να μιλήσω για του Κούρδου στη Συρία, κυρίω στα πλαίσια της, των σειράξεων στη Μέση Ανατολή και να δείξω ποιε είναι συνέπειε τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ηθαγένεια για του απάτριδε βάσει στι διάφορε προκλήσει που εντοπίζονται στη μελέτη που διαβάστηκε προηγουμένως. Θα ήθελα να τονίσω και συμπληρωματική προοπτική που νομίζω ότι θα πρέπει να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αξιολογεί την πολιτική που ακολουθεί για την ανηθαγένεια και σχετίζεται με τη διπλή πρόκληση. Δηλαδή να είναι κανείς χωρίς πατρίδα και να είναι ένας λαός με ανηθαγένεια που αυτό ισχύει για πάρα πολλούς Κούρδους. Ε, η ανηθαγένεια είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όχι μόνο αυτό. Ένα ισχυρό επιχείρημα που αναφέρεται και στη μελέτη τη Δόκτωρος Βαν είναι ότι η ανιθαγένεια γίνεται, είναι προϊόν παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι και αίτιο άλλων προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραδείγματο χάρη, στην περίπτωση των Κούρδων στη Συρία, η περιθωριοποίηση οδήγησε σε διακριτική δημογραφική έρευνα που τελικά κατέληξαν να γίνουν μια ανοιχτή ε, ανιθαγενής οι Κούρδοι στην απογραφή. Λοιπόν, στο διάταγμα 49 κάποιοι ε, Κούρδοι ε, μετρήθηκαν, διπλασιάστηκε ο αριθμός των ε, Κούρδων και έγινε, ήταν διάκριση που έγινε μέσω του νόμου ψηφίστηκε. Και τελικά η ηθαγένεια πέρασε από τους γονείς στα παιδιά μέσα από τα λάθη που έγιναν. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι Κούρδοι τελικά ε, έγιναν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες ατόμων με το πρόβλημα της ελλείψης ηθαγένειας και αν ηθαγενείς Κούρδοι στη Συρία επέφεραν από διάφορες παραδείγματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναφέρομαι μόνο σε δικαιώματα δικαιώματα ψήφου, παραδείγματο χάρη, συμμετοχή σε κυβέρνηση, όχι μόνο αυτά όμω, και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στερούνται. Όπω πρόσβαση σε κρατική εκπαίδευση, επίσημη απασχόληση, πρόσβαση σε έγγραφα, ε, ακόμα και θέματα προσωπικής ασφαλείας εθίδιοντο. Όπως προανέφερα, το διάταγμα 49 που εισήχθη το 2011 και κατήργησε την, ε, τελικά ε, την επικότητα που είχαν κάποιοι Κούρδοι. μάλιστα κατήργησε το καθεστώς απάτητος για τους Κούρδους. Ήταν θετικό βήμα, οι λόγοι ήταν πολιτικοί περισσότερο παρά ανθρωπιστικοί και πολλοί από τους πρόσφυγες, τους Κούρδους που εκτοπίστηκαν από τη Συρία λόγω της κρίσεως της τωρινής ήταν απάτηδες πριν φύγουν και τώρα δεν έχουν υπηκότητα στην εξορία τους και το πρόβλημα προκύπτει εκεί. Τι θα συμβεί όταν τελικά θα μπορέσουν να επιστρέψουν, θα μπορέσουν να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, ακόμα και εκείνοι που θεωρητικά έχουν ωφεληθεί από το διάταγμα που ψηφίστηκε το 2011, ακόμα αισθάνονται τις συνέπειες ε, δεν έχουν ωφεληθεί ακόμα διότι η σύγκρουση έχει διαταράξει την ομαλότητα. Ακόμα και το δικαίωμα της ζωής απειλείται. Οπότε έρχομαι στο δεύτερο ζήτημα που ήθελα να υπογραμμίσω και που δεν έφυγε στη μελέτη της δόκτωρος Βαμβάς. Δηλαδή της ανιθαγένειας των λαών. Πέρα του να έχει υποφέρει κανείς από τις συνέπειες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, λόγω ανιθαγένειας, λόγω της είναι ο μεγαλύτερος αν ανιθαγενής λαός οι Κούρδοι. Δεν έχουν χώρα, δεν ελέγχουν πολιτικά την πατρίδα τους, τις περιοχές που θεωρούνται πατρίδα τους και δεν συμμετέχουν επίσημα, ούτε εντάσσονται επίσημα, ούτε έχουν ίσες οικονομικές ευκαιρίες στις χώρες που καλύπτουν το λεγόμενο Κουρδιστάν. Στην περίπτωση λοιπόν των απάτηδων Κούρδων στη Συρία και άλλων, η απόκτηση της ηθαγένειας ίσως να μην αρκεί για να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανηθαγένεια όπως είναι η πλήρη συμμετοχή σε πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή. Εν γέννη λοιπόν η ανηθαγένεια έχει και με τις δύο έννοιες διαπιστώνεται εδώ. Αισθάνονται αποκλεισμένοι άνθρωποι και αισθάνονται ότι δεν ανήκουν κάπου, του λείπει ταυτότητα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κοινωνικέ συγκρούσει. Μπορεί να ειδωθεί και σε ένα θέμα που αφορά και τη μετανάστευση. Δηλαδή, οι κοινότητε τη διασπορά πολύ συχνά αισθάνονται μια μόνιμη ανασφάλεια σε όποια χώρα και να ζουν, παρόλο που τους έχει δοθεί υπηκοότητα και έχουν κοινωνική, κοινωνικά εργετήματα και λοιπά και παιδεία, αισθάνονται ότι δεν έχουν πατρίδα και ίσως χρειάζεται γενιές τελικά για να εξαλειφθεί αυτό το συνέστημα. Όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όσον αφορά την ανηθαγένεια είναι θετικό να σημειώσουμε ότι οι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ενώσης έχουν συμπεριλάβει δράσει που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο θέμα, όμω κάτι που αναφέρεται και στην έκθεση, φαίνεται λέγω ότι χρειάζεται πιο συγκεκριμένη συντονισμένη δράση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανηθαγένειας και λαμβάνοντας υπόψη και ότι η ανηθαγένεια είναι ένα πρόβλημα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που όμως επηρεάζει σειρά προτεραιοτήτων που έχει θέσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις προτεραιότητες κατά χώρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρονται στην έκθεση της κυρίας Βαμβάς, ε, έχουμε τη Συρία και χώρες που πλήττονται από τη σύγκρουση όπως είναι το Ιράκ. Και άλλη πρόκληση, άλλο πρόβλημα που μπορεί να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν σχεδιάζει μια απάντηση όσον αφορά την ανιθαγένεια σε σχέση με τις συγκρούσεις. Σχετίζεται με την de facto ανιθαγένεια. Σε πρόσφατη επίσκεψη στο Ιράκ, συνάντησα ένα επιβιώσοντα από το Σιντζάρ, είχε χάσει τα πάντα, όλα τα υπάρχοντά του, περιουσία, ταυτότητες, τα πάντα και για λόγου ασφαλεία δεν μπορούσε να επιστρέψει, δεν μπορούσε να πάει στη Βαγδάτη και να βγάλει νέα έγγραφα. Και είχε πρόβλημα λοιπόν να, ε, να απολαύσει τα δικαιώματα του εκείνου πολίτου και να του προσφερθούν υπηρεσίε. Και είπε και παραθέτω, η ταυτότητά μου ε, διαγράφηκε. Όλα τα έγγραφα τα έκαψε το Ισλαμικό κράτος. Δεν έχω πλέον ιστορία, δεν έχει αξία η ύπαρξή μου. Ε, Κλείνοντα, θεωρώ σημαντικό να τονίσουμε ότι η ανηθαγένεια είναι ανθρωπογενής Άρα μπορεί να επιληθεί σαν πρόβλημα από τη στιγμή που υπάρξει κατανόηση και προθυμία για την αντιμετώπιση των αιτίων. Και έκθεση της δόκτωρος Βαμβάς και αυτή η ανταλλαγή των απόψεων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συνεπώς είναι πολύ ευπρόσδεκτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γκριν. Τώρα έχω προβλέψει να, να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάρετ Ομπράιαν, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ή μάλλον όχι. Μετά που θα μιλήσουν τα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Λοκμήλη πρώτα. Thank you, uh, Chair, and thank Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την υπέροχη αυτή μελέτη. Είναι πολύ καλό να ακούει κανείς και να μαθαίνει τόσα πράγματα. Νομίζω ότι η ομάδα των Πρασίνων ξεκίνησε την όλη προσπάθεια. Όλοι μας όμως θα πρέπει να δούμε ότι δίδεται κάποια συνέχεια. Λέτε ότι 80% των ανθρώπων ότι λείπει, οφείλεται το πρόβλημα στην έλλειψη πολιτικής βούλησης. Αν δούμε τις χώρες που δεν επικύρωσαν την σύμβαση του 1994, έχουμε την Κύπρο, Εσθονία, Γαλλία, α, συγγνώμη, Κύπρος, Εσθονία, Μάλτα και Πολωνία. Δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή και μετά έχουμε τη σύμβαση του 61 για την μείωση του προβλήματος ανιθαγένειας. Δεν έχει επιβληθεί την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, Πολωνία, Σλοβανία, Ισπανία και μια-δυο άλλες χώρες. Καλύπτουν το 80% που αναφέρατε για το πρόβλημα υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Στη μελέτη λέει ότι στη η Γερμανία μου έχει... η χώρα μου έχει κυρώσει τη σύμβαση. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Θα μπορούσατε να δώσετε λεπτομέρειες. Και μετά ίσως θα αναφερθεί στο θέμα υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Του θέτω το ερώτημα. Είπατε ότι είπατε αρμοστία το ΙΕ. Κάνει μια εκστρατεία για να λήξει το πρόβλημα τη ανηθαγένεια μέχρι το 2024. Πόσο το προωθεί το θέμα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης στα διάφορα πολυμερή βήματα συζητήσεων και πρακτικό θέμα και σύσταση. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης μήπως μπορούσε να συμπεριλάβει κάποιες δράσεις στο σχέδιο δράσης και να βρει, να ετοιμάσει μια εργαλειοθήκη ευρωπαϊκή για την καταπολέμηση του προβλήματος. Εξέλαβα από αυτά που είπατε ότι στη μελέτη μελετήσατε διάφορες χώρες και βάλατε μια μάρα κτήρ φαντοστού, Συρία, δημο, ε, Δομινικανή, Δημοκρατία, ε, ίσως η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα μπορούσε να μας πει τι κάνουμε για τις συγκεκριμένες χώρες. Ο κύριος Παντζέρη κινείται και εργάζεται για μια ετήσια έκθεση που έχουμε αν συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό θέμα θα μπορούμε να συνεργαστούμε ίσως και να ετοιμάσουμε μια παράγραφο για το πρόβλημα που συζητάμε για την ανηθαγένεια. Δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί κάποια πρόταση έχει ο κ. Μάνλη να ζητήσουμε κάποιο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το πρόβλημα της ανηθαγένειας. Ίσως η Επιτροπή μας θα μπορούσε να το ζητήσει αυτό. Η κυρία Πόστ, ή το λόγο. Βρήκα πάρα πολύ ενημερωτική τη συζήτηση, πολύ ε, επικοδομητικές απόψεις και σκέφτηκα αρκετά θέματα που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Σκέφτηκα, ας πούμε, τον χάρτη μας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που ο χάρτης αυτός δεν αναφέρεται στο δικαίωμα στην ανιθαγένεια, στην ε, σύμβαση αναφέρεται ότι οι ανηθαγενείς ε, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτων χωρών. Εκείνο όμως που λείπει στη μελέτη και αυτό είναι και το ερώτημά μου είναι το εξής. Στη μελέτη σας ήρθατε σε επαφή με ανηθαγενείς Ρωμά. Ξέρω ότι υπάρχουν υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου Υπάρχουν ε, πολλές κοινότητες ε, Ρωμά. Κατοντάδες χιλιάδες ε, Ρωμά είναι ανιταγενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τον αριθμό γνωρίζω εγώ. Αυτοί όλοι είναι διάσπαρτοι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να σας πω ότι με εκπλήσει λιγάκι η κατάσταση γιατί πρόκειται για μια ξεκάθαρη υπόθεση και αυτό ε, διατρέχει πολλές γενναίες και ούτε καν λόγος δεν γίνεται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί αυτό το ερώτημα ούτε καν τίγεται. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση ε, αποτελεί κατάφορη διάκριση εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Έγινε λόγος ε, για τη Σερβία από ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, έγινε, έγιναν κάποιες συζητήσεις με γυναίκες Ρωμά που δεν μπορούν ούτε καν να γεννήσουν τα παιδιά τους στα νοσοκομεία, ούτε καν να θαυτούν στα νεκροταφεία. Αυτά συμβαίνουν εδώ μπροστά στην πόρτα μας και νομίζω ότι θα πρέπει να τα θίξουμε. Πρέπει να σας πω ότι έχω γράψει πάρα πολλές προτάσεις, έχω και άλλα ερωτήματα να θέσω που θα μου επιτρέψετε να τα θέσω αργότερα. Πρόκειται ας πούμε και για τη συνεργασία με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ίσως και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μπορούμε κάτι να κάνουμε. Πάντως ε, αυτό το θέμα, το θέμα της εμπορίας ανθρώπων, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το ερώτημά μου λοιπόν, και θα το επαναλάβω, ξέρετε κάτι σχετικά με την κατάσταση των Ρωμά και γιατί δεν θίγεται καθόλου το θέμα των Ρωμά στη μελέτη σας και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Γιατί όπως σας είπα αυτό γίνεται στα μάτια μας, μπροστά μας, μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Sí, señora Post, muchas gracias. Έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Πόστε, ε, ο κύριος Αστραβίτσιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη σελίδα 22 η μελέτη λέει το εξής. Η ανιθαγένεια δεν είναι προτεραιότητα ρητός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έστω, μέχρι εδώ το καταλαβαίνω. Ωστόσο, η άνηθαγενείς και μάλιστα στις ε, γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο πιθανό να θέλουν να μεταναστεύσουν και να βρουν αλλού να ζήσουν. Γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και η μετανάστευση είναι προτεραιότητα, είναι γραμμή πολιτική γραμμή υψηλής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λογική σύνδεση μεταξύ των δύο, δηλαδή η ανηθαγένεια θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από τη στιγμή που δημιουργεί μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση. Έτσι δεν είναι. Καλά δεν τα λέω. Thank you very much. Mr. Ja, dank u wel. Dank u aan alle leden van, van het panel voor de interessante... Ο κύριο Ντέμεν Σμέκερ. Ε, σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσε συνεισφορέ συνεισφορές Η κατάσταση στη Συρία και στο Ιράκ είναι γνωστή δεν βελτιώνεται η κατάσταση των ανιθαγενών σε αυτές τις χώρες. Η κρίση στη Συρία και στο Ιράκ έχει επιδεινώσει την κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους, άρα το πρόβλημα οξύνεται. Επομένως, όντως θα πρέπει η ανηθαγένεια να είναι προτεραιότητά μας. Και σε, σε αυτό που είπε η κυρία Φαμπάστ παρατήρησα και το εξής. Είπε ότι δύο από τις χώρες ε, που είναι μέσα στις δέκα πρώτες είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ σωστά υπογράμμισε το συσχετισμό μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης. Επομένως, ρωτώ, μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε ασχολούμενοι με το πρόβλημα αυτό εντός των ευρωπαϊκών συνόρων για να μην πλήτεται η αξιοπιστία μας. Πώς μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι έναντι του υπολείπου κόσμου εάν δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πώς θα είμαστε αξιόπιστοι έναντι των τρίτων χωρών όταν Δύο χώρες από τις δέκα πρώτες είναι κράτη ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα πρώτες εννοώ ως προς τον αριθμό των ανηθαγενών. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον αριθμό των ανηθαγενών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ενδείξεις ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Ε, τι, μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Muchas gracias, señor Voy a dar la palabra ahora ya sí al señor Garrett O'Brien, eh, que también ha recibido. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Γκάρετ Ομπράιαν. Έχετε δεχτεί ερώτηση από τους βουλευτές, παρακαλώ. Very much. Um... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω καλωσορίζοντας τη χρησιμότατη πληρέστατη έκθεση και τις εμπεριεχόμενες συστάσεις προς την εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Σωστά σημειώνεται ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική για την ανηθαγένεια για την ώρα. Πολλά όμως γίνονται στα πλαίσια προσπαθειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα παιδιών, ισότητα των φύλων και αποφυγή συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει την ηθαγένεια σε πολλές στοιχείες της εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών σχέσεων, στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας και στις διαδικασίες της διευρύνσεως. Η ανηθαγένεια εντοπίστηκε ως προτεραιότητα τις στρατηγικές καταχώρε και τα ανθρώπινα δικαιώματα για διάφορε χώρε με σημαντικά προβλήματα ανηθαγένεια και τα θέτουμε στη συζήτηση με τι κυβερνήσει αυτέ Σημαντικά προβλήματα ανιθαγένειας ήδη έχουν εντοπιστεί και αναφερθεί σε επισκέψει υψηλού επίπεδου και σε δημόσιε δηλώσει τα τελευταία χρόνια. Πιο το παράδειγμα ίσω είναι το Μιανμάρ όπου συνεχώς αναφερόμαστε στην κατάσταση των Ροχίνγκα σε διμερείς ε, δηλώσεις, επισκέψεις ε, και στη συζητήση σε πολυμερή βήματα συζητήσεων. Επιπροσθέτως, όπως σημαίνεται στην έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί διάφορα προγράμματα για την υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων. Πολλά από αυτά συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα που σχετίζονται με, τους, ε, με τα προβλήματα σαν και εκτατική χρηματοδότησης για UNICEF, ONRWA, τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και υποστηρίζουμε ε, τους διάφορους φορείς που κινούνται για το πολέμηση του φαινομένου. πράγματος για αντιμετωπιστεί κρίση των προσφύγων από τη Συρία. Η Στατική Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεργασία με τρίτε χώρε στον τομέα τη μετανάστευση και του ασύλου εντοπίζει την ανηθαγένεια σαν βασικό στόχο, βασική προτεραιότητα Επίση, παρέχουμε στήριξη σε οργανώσεις κοινωνία των πολιτών για τη δουλειά που κάνουν όσον αφορά την ανιθαγένεια. 1,6 εκατομμύρια ευρώ διατέθησαν σε προγράμματα για την ανιθαγένεια τελευταία τριετία συμπεριλαμβανομένου ενό προγράμματο που περιγράφει πρόσφατα για την υποστήριξη τη ομαλοποίηση των επικών τη Δομινικανή Δημοκρατία με ε, καταγωγή από την ΑΕΤ. Έχουμε εντοπίσει σε προτάσει την ανιθαγένεια σαν στόχο και 5 εκατομμύρια έχουν διτεθεί για προγράμματα για μετανάστευση και ανιθαγένεια. Η ανιθαγένεια επίση έχει εντοπιστεί σαν βασική πρόκληση στη διεύρυνση, κυρίω όσον αφορά του ανιθαγενεί Ρωμά των Δυτικών Βαλκανίων και χρηματοδοτούμε διάφορα προγράμματα ανιθαγένεια στην εν περιοχή. Κάποια τα προγράμματα εφαρμόζονται από την Υποτερμοστία του ΟΗΕ για τι πρόσφυγε. Τώρα αναπτύσσουμε ένα πλαίσιο πλαίσιο για που θα θέτουμε τα θέματα ανηθαγενεία σε σχέση με τρίτε χώρε. Ήταν δέσμευση που ανελήφθη στο σχέδιο δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Έχουμε συνεργαστεί στενά με την ύπατη αρμοστία για τι πρόσφυγε του ΟΗΕ. Εντοπίσαμε διάφορε χώρε που έχουν προτεραιότητα, βασικά μηνύματα που πρέπει να στείλουμε. Και είναι ένα εργοτάξιο για την ώρα, αλλά θα προχωρήσουμε τον επόμενο χρόνο. Πρόθεσή μα ήταν να συμπληρώσουμε την στη δουλειά που κάνει η πατερμοστία για τι πρόσφυγε του ΟΗΕ, προωθώντα το ζήτημα θα ζητήσουμε στις προσωπίες μας να συνεργαστούμε με τους ομολόγους στο τσίπα της του ΟΗΕ όταν θα εφαρμόζουν τα εν μέτρα. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι κάνουμε σε κάθε χώρα που εντοπίζεται στην έκθεσή σας. Το μόνο που θα πω είναι ότι σίγουρα στην περίπτωση των Μιγκανής Δημοκρατίας και το Μιανμάρ ε, ήταν θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε θέσει επανειλημμένα σε επαφές με τις αρχές των χωρών αυτών και όπως προανέφερα επίσης χρηματοδοτούμε δραστηριότητε που καταπολεμούν το πρόβλημα τη ανηθαγένεια και σε σχέση με την κρίση στη Συρία, πάρα πολύ προσοχή δίδεται στο όλο θέμα. Πράγματι, στο μέτρο του δυνατού θέλουμε να στηρίξουμε την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ στην εκστρατεία που διεξαγάγει συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου που ελπίζουμε να ολοκληρωθεί τάχιστα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ομπράιν. Τέλος, να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους για δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Φαμπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέροντα και χρήσιμα τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι κάποιες ερωτήσεις ήδη απαντήθηκαν, κάποια θέματα ήδη καλύφθηκαν. Θα ήθελα απλώς να θίξω δύο σημεία. Το πρώτο που αφορά την έλλειψη της προσοχής όσον αφορά την κατάσταση των ανιθαγενών Ρώμα εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στα δικαιώματα, με την πρόσβαση σε κάποια είδη εγγράφων για τους Ρωμά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν περιπτώσεις ανιθαγένειας μεταξύ αυτών, όμως η τεράστια πλειοψηφία των Ρωμά που ζουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών αυτής, αναγνωρίζονται ως υπήκοοι των χωρών Οπότε τα προβλήματα δεν θα πρέπει να ειδωθούν απαραίτητα σαν προβλήματα ανηθαγένεια, αυτά καθε αυτά, αλλά σαν ευρύτερα προβλήματα που άπτονται τη πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί που διαφέρουν τα πράγματα κάπω είναι κυρίω στι χώρε τη πρώην Ιουγκοσλαβία, όπου υπάρχουν πραγματικά προβλήματα όσον αφορά τη μην αναγνώριση υπηκότητα για κάποιε ομάδε Ρωμά μετά την, τον διαμελισμό τη Ιουγκοσλαβία. Θα ήθελα μετά να πω και κάτι σχετικά με το θέμα το 80% πολιτική βούληση, 20% τεχνική, τεχνογνωσία. Νομίζω ότι κάποια σχόλια που ακούστηκαν εδώ σήμερα και κάποιες από τις συστάσεις που αναφέρονται στην έκθεση έχουν στόχο ακριβώς το βασικό θέμα της ορατότητας για το πρόβλημα. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά συζητώντας τουλάχιστον το θέμα της πολιτικής βουλήσεως αν η ηθαγένεια τίθεται σαν πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο σε σχέση με άλλα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά σαν ένα συγκεκριμένο, συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλωσορίζω θερμά τις ευκαιρίες που δημιουργούνται να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα ασχολείται με το θέμα να γίνονται καταγγελίες για προβλήματα ανηθαγένειας στις αιτήσεις εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι θα κατανοηθεί καλύτερα το πρόβλημα, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για έλεγχο των χωρών εκείνων που χρειάζεται μεταρρύθμιση, να λογοδοτήσουν αυτέ οι χώρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάνιγκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και για τα σχόλιά σας και εγώ ακροθυγώς θα αναφερθώ στο θέμα της πολιτικής βούλησης. Κοιτάξτε σίγουρα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει θέμα αδράνειας. Αυτές οι συμβάσεις υπήρχαν επιμακρών και σε πολλές περιπτώσεις μόλις πρόσφατα τα κράτη-μέλη είδαν με σοβαρότητα ε, τις συμβάσεις και είδαν τι αξία έχουν και το πώς μπορούν να εξασφαλίσουν καλή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σφαιρικά και το ρόλο που μπορεί να παίξει κάθε κράτος μέλος στηρίζοντας την προσπάθεια εξάλληψης του φαινομένου της ανιθαγένειας ε, συμμετέχοντας, προσχωρώντας στις δύο συμβάσεις. Γιατί λέω ότι είναι θέμα αδράνειας. Οι, οι νόμοι της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας για την υπηκότητα είναι πάρα πολύ καλοί και αν εφαρμοστούν σωστά αυτοί οι νόμοι δεν δημιουργούν πρόβλημα ανηθαγένειας. Όμως καμία από τις χώρες δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του 1961 για τη μείωση της ανηθαγένειας. Άρα δεν υπάρχει εμπόδιο όσον αφορά το εθνικό δίκαιο. Είναι θέμα ε, εκ του εκτελεστικού κλάδου και νομοθετικού κλάδου, οι δύο κλάδοι να καθίσουν και να εξετάσουν σοβαρά και να δουν το θέμα της προσχώρησης. Με τα χαρά στην Ιταλία τουλάχιστον το Συμβούλιο των Υπουργών έχει εγκρίνει την προσχώρηση της Ιταλίας. Ε, κινούνται γρήγορα και τα πράγματα. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι και το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε στα πλαίσια μη συνεδρία υψηλού επίπεδου για το κράτο δικαίου στον ΟΗΕ το 2012 ότι όλα τα κράτη-μέλη θα κυρώσουν ή θα προσχωρήσουν στην σύμβαση του 1954 που αφορά το καθεστώ των ανηθαγενών. Έχουμε τέσσερις χώρες που δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο όπως αναφέρει και Εστονία, Πολωνία, Μάλτα και Κύπρος. Τώρα, όσον αφορά το συναφές θέμα, δηλαδή αν αντιμετώπιση του προβλήματος εντός των σειρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι κάτι σημαντικό, σίγουρα είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορούν να ηγηθούν, να δώσουν το παράδειγμα. Και σίγουρα η προσχώρηση στη, στη σύμβαση δείχνει ότι μπορούν να ηγηθούν στο παγκόσμιο προσκήνιο. Άλλο τρόπος να εξασφαλίσουμε τη μείωση των ενθαγενών ατόμων. Αυτό χρειάζεται μεταρρύθμιση νομοθεσιών περί ηθαγενεία. Με τα χαρά λέω ότι σήμερα το Εστονικό Κοινοβούλιο ψήφισε μεταρρύθμιση του νόμου περί ηθαγένεια και εκεί προβλέπεται ότι η απόκτηση υπηκότητα από του ανηθαγενεί διευκολύνεται και τα παιδιά που γεννήθηκαν από γονεί, ανηθαγενεί αυτομάτω αποκτούν υπηκότητα. Δεν πρέπει να κάνουν κάποια δήλωση οι γονεί Τέτοιου είδου βήματα απαιτούνται σε χώρες που έχουν ε, ε, προβλήματα. Αν περισσότερες χώρες κάνουν αυτό το πράγμα και διευκολυνθεί η απόκτηση υπηκότητας, θα μειωθούν οι αριθμοί των ηθαγενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε αυτό να γίνει πιο γρήγορα. Τέλος. Όσον αφορά τα κίνητρα για τη μετανάστευση, δεν νομίζω ότι είναι ηθαγένεια είναι κίνητρο για μετανάστευση. Δίνει ένα πρόξιμο αν τους αρνούνται ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα που γεννήθηκαν και γεννήθηκαν οι γονεί του, είναι πολύ πιθανό να μπουν στο πλοίο ή να κάνουν πολύ επικίνδυνα ταξίδια τα πάντων άνθρωποι, να κάνουν το γύρο του κόσμου για να βρουν κάπου προστασία σαν πρόσφυγε. Αυτό είναι γεγονό. Θα πρέπει να κρυζώσουμε το πρόβλημα για του πρόσφυγε. Ε, ένα από τα αίτια είναι η ανιθαγένεια. Δεν είναι σύμπτωση ότι η πατιαμοστία για του πρόσφυγε πήρε την ευθύνη να αντιμετωπίσει την ανιθαγένεια το 1994. Αποτέλεσμα ψηφίσματο Γενική Συνελεύσεω λόγω τη διάλυση τη Σοβιετική Ενώσεω, πριν από μερικά χρόνια και του διαμελισμού τη Ιουγκοσλαβία. Τα δύο γεγονότα αυτά δημιούργησαν τεράστιου αριθμού ανιθαγενών και τεράστιε μετακινήσει πληθυσμών κόσμου που έψαχνε προστασία ω πρόσφυγε, συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων που κατέφθασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προ όφελο όλων των χωρών να επιλύσουν το πρόβλημα και έτσι να εκκριζώσουν ένα από τα αίτια της ανηθαγένειας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Μάνλη κύριε Αμπτελσαλάμ. Για δύο λεπτά, για να εξάγουμε τα τελικά μας συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θέλω να θίξω είναι το θέμα της ε, Συρίας και των ε, προεκτάσεων, κυρίως σε σχέση με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Οι Παλαιστίνοι βρίσκονται στη Συρία εδώ και 67 χρόνια και έχουμε περίπου 50.000 ε, Παλαιστίνιους πρόσφυγες που βρίσκονται στη Συρία και λόγω των φρικαλαιοτήτων του πολέμου είναι αναγκασμένοι να φύγουν στο εξωτερικό. Έχουν προβλήματα και νομικής φύσεως. Ο Λιβανός δεν τους αντιμετωπίζει καν ως πρόσφυγες. Άρα δηλαδή η δική τους κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και αυτό που χρειάζεται εδώ είναι μια στεναρή στάση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Λίβανο του στέλνει πίσω και αυτοί πεθαίνουν στη Συρία. Αυτό είχα να πω ως κατακλείδα της παρέμβασής μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Γκριν έχει το λόγο. Κοιτάξτε, το, η αντιμετώπιση της ανιθαγένειας ε, και η προστασία των μειονοτήτων ε, σε χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς επιθυμούμε το θέμα αυτό να επιληθεί ως προτεραιότητα όσον αφορά τα, ε, τις ανησυχίες Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Πόστη θα πει κάτι και μετά η κυρία Βανβάστ. Παρακαλώ. Νομίζω ότι με παρεξηγήσατε, δηλαδή όταν εγώ μίλησα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μίλησα για εκατοντάδες χιλιάδες, δεν εννοούσα τους Ρωμά. Μιλούσα ιδιαίτερα για τους ανιθαγενείς Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και βεβαίως και στην πρώην Ιουγκοσλαβία και για τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στους Ρωμά που διέφυγαν λόγω των ε, Βαλκανικών πολέμων. Απλά ε, να το σημειώσετε αυτό ότι όταν μίλησα προηγουμένως για τους Ρωμά δεν εννοούσα γενικότερα τους Ρωμά που πίστανται διακρίσεις αλλά τους ανιθαγενείς Ρωμά. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, δώσαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι είχαμε προβλέψει. Είναι όμως ένα σημαντικό ζήτημα, ένα νέο ζήτημα η κατάσταση των ανήθαγενών στον κόσμο και γι' αυτό είναι καλό το, το γεγονός ότι το ανοίξαμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους συμμετέχοντες. του καθενός και της κάθε μία σας ξεχωριστά. Εκ μέρους του ε, ΡΑΕΙΦ σας ευχαριστώ θερμά, ειδικότερα από τότε που ξεκίνησε ε, το μαστίγωμα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες. Ελπίζαμε ότι η σύζυγός του θα ήταν σε θέση να μας μιλήσει ε, σήμερα το απόγευμα. Τεχνικώς δεν είναι αυτό εφικτό. Είναι δύο τα βίντεο που, θα θέλ, που θέλουμε να σας δείξουμε. Θα σας τα δείξω λοιπόν και μετά θα σας ενημερώσω για την κατάσταση. Το πρώτο βίντεο το γυρίσαμε με την οικογένεια Ατού, η οποία βρίσκεται σε εξορία στον Καναδά αυτή τη στιγμή, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι μέρος του μαραθωνίου της Διεθνούς Αμνηστίας, ε, της δράσης που κάνουμε κάθε Δεκέμβριο το right for right, γράψε για ένα δικαίωμα. Επομένως έχουμε σύνταξη επιστολής γιατί είναι μέρος της δράσης μας αυτής. Και το δεύτερο είναι ένα μήνυμα από βίντεο ε, από τη γυναίκα του στον Καναδά, το οποίο είναι ε, στα γαλλικά, θα υπάρχει μετάφραση από τους δερμηνείς. Επομένως σας ε, δείχνουμε το βίντεο και μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μετάφραση. for Όσο περιμένουμε τα βίντεο να σας ενημερώσω για την κατάσταση, ο Ραΐφ Μπατάουι καταδικάστηκε πέρσι σε 10 χρόνια φυλάκιση και σε χίλιες βουρδουλιές έχει, διότι δημιούργησε ένα blog διαδικτυακό στο οποίο ενθάρρυνε άτομα από τη Σαουδική Αραβία να εκφράσουν τις απόψεις τους για την πολιτική και δημόσια σφαίρα. Ε, στις 9 Ιανουαρίου Παρασκευή πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησε το μαστίγωμα ε, του έδωσαν 50 μαστιγώματα ε, από τα χίλια 50 λοιπόν κάθε Παρασκευή μπροστά στο ε, τέμενο στο ιερό στη Τζέντα ε, με κοινό. Αυτή είναι η ποινή του. Κάθε Παρασκευή λοιπόν 50 βουρδουλιές. Ε, δόθηκε μεγάλη προσοχή στο θέμα από κυβερνήσεις, ε, το διεθνή τύπο την περασμένη Παρασκευή θα, ε, είχε πάλι τις 50 βουρδουλιές έξω από το τέμενο της Τζέντα. Αυτό δεν έγινε την περασμένη Παρασκευή γιατί ε, την ώρα που τον οδηγούσαν ο γιατρός τον εξέτασε και είπε ότι οι βουρδουλιές δεν είχαν αρκετά θεραπευθεί για να μπορέσει να αντέξει τις επόμενες 50. Άρα τις μετέθεσαν για αυτήν εδώ την Παρασκευή και ε, μεθαύριο Παρασκευή θα ε, του δώσουν αυτές τις 50 βουρδουλές το δεύτερη, τη δεύτερη δόση αν θέλετε γιατί έχουν περάσει δύο εβδομάδες και θα έχουν θεραπευθεί αρκετά οι πρώτες 50. Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η εκστρατεία υπεράσπισης του. Η υπόθεση πήγε στο ανώτατο δικαστήριο πριν τα Χριστούγεννα το Δεκέμβριο. Αυτό είναι μέτρο ρουτίνας και όχι ε, και όχι ως αποτέλεσμα της διεθνούς πίεσης. Επομένως δεν τρέχουμε και πάρα πολλές ελπίδες ότι την Παρασκευή δεν θα ε, δοθούν αυτές οι βουρδουλές. Δεν ξέρω τώρα αν έχει ε, αποκατασταθεί η βλάβη τεχνική και μπορούμε να δούμε τα βίντεο. Λοιπόν,

Eh, λοιπόν, δεν υπάρχει ήχος. Θα διαβάσω εγώ το κείμενο ε, της συζύγου του Ραΐφ Μπαντάουι. Οι διερμηνείς έχουν το κείμενο και βεβαίως μπορούν να το μεταφράσουν. Είμαι η Ενσάφ Χαϊντάρ, η γυναίκα του Ραΐφ Μπαντάουι. Ο Ραΐφ είναι ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδρυτής του ε, φιλελεύθερου δικτύου της Σαουδικής Αραβίας. Είναι κρατούμενος για τις απόψεις τους στο βασίλειο του διαλόγου των θρησκειών. Είναι ένας άνθρωπος απλός, ειρηνικός, εξαιρετικός σύζυγος, τρυφερός πατέρας. Τα γραπτά του ασχολούνται με διάφορα θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, τις πολιτικές ελευθερίες, τις θρησκευτικέ ελευθερίες. Μία από τις παραθέσεις, ε, τις πιο σημαντικές ε, του Ραΐφ είναι και η εξή και παραθέτω. Επιθυμώ τη ζωή ε, για όλους αυτούς οι οποίοι θέλησαν το δικό μου θάνατο. Επιθυμώ τον, τη λογική ε, σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλησαν να με θεωρήσουν εμένα ως ε, αδαή η πίεση που ασκείται από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αποτελεσματική ε, λόγω του βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμά για τη θέση που υιοθετείτε και ε, θα ήθελα να συνεχίσετε να έχετε αυτή τη θέση και να συνεχίσετε να ασκείτε αυτή την πίεση μέχρι να ελευθερωθεί ο Ραΐφ. Ευχαριστώ. Αυτά είναι λοιπόν τα λόγια της Ενσάφ Χαϊντάρ, της συζύγου της Ραΐφ Πανταουή. Ε, έρχομαι τώρα και διαβάζω το γράμμα του παιδιού του Ραΐφ Πανταουή πλαίσιο της εκστρατείας Right for Rights. Ε, πατέρα πίστεψέ με, ποτέ δεν πίστεψα ότι θα ζούσα χωρίς ε, εσένα. Ποτέ δεν, ποτέ δεν, είχα, δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι δεν θα με ξυπνούσε κάθε πρωί για να πάω στο σχολείο όπω συνήθω. Ποτέ δεν φανταζόμουν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Είσαι στη φυλακή μακριά μου γιατί αγωνίστηκε για τι ιδέε σου. Είσαι ένα άνθρωπο ειρηνικό που αγαπάει τον κόσμο και επιθυμεί όλο ο κόσμο να του συμβαίνουν καλά πράγματα. Γιατί είσαι στη φυλακή, αυτό το ερώτημα θέτω στον εαυτό μου κάθε μέρα. Είναι αλήθεια ότι είσαι στη φυλακή γιατί έφτιαξε μια ιστοσελίδα που ενθαρρύνει τον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο. Όταν η μαμά είπε ότι ήσουν στη φυλακή λόγω των ιδεών σου, έψαξα το όνομά σου στο Google και με έκπληξη είδα τη στήριξη την οποία ε, ε, δέχεσαι από όλο τον κόσμο. Χωρί τη μαμά θα είχαμε υποφέρει ακόμα περισσότερο από την αποσία σου. Η μαμά είναι δυνατή, μην ανησυχεί. Δυόμιση χρόνια τώρα ε, κάνει ό,τι μπορεί για να αντισταθμίσει την αποσία σου, αλλά τίποτα δεν μπορεί να, να σε αντικαταστήσει. Οι αδερφέ μου και εγώ ε, αναρωτιόμαστε κρυφά ε, πώς θα μπορούσαμε να σε κάνουμε να βγει από τη φυλακή. Η Μίριαμ είπε ότι θα πήγαινε στην Σαουδική Αραβία, ότι θα ε, ε έσπαγε τους τοίχους της φυλακής και θα χτυπούσε του φρουρού για να βγει ο μπαμπά από τη φυλακή πρέπει ο μπαμπάς να επιστρέψει στο σπίτι. Περιμένουμε τη μέρα όπου το, το αεροπλάνο θα έρθει στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, θα με δεις να περιμένω, ε, δεν θα σταματήσω μέχρι ότου να με πάρει στα χέρια σου, να με πάρει αγκαλιά και να στεγνώσει τα δάκρυα άμμου. Ε, ο Ντουντή ο θησαυρό σου. Αυτό είναι το τέλος λοιπόν του γράμματο του παιδιού του Ραϊφ Μπανταουή. Ο κ. Νίκος παίρνει το λόγο και λέει ότι... Ε, οι αρχές ασχολούνται ήδη βεβαίως και γνωρίζουν ότι το θέμα αυτό βρίσκεται στη διεθνή επικαιρότητα, γνωρίζουν ότι δεν δίνεται καλή εντύπωση για τη Σαουδική Αραβία στον υπόλοιπο κόσμο και θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να ακούσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να της λέει ότι αυτό αποτελεί σοβαρή ε, παράβαση διεθνούς δικαίου. Είναι κάτι το οποίο έχει πει ξεκάθαρα και ο υπατσαρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άρα αυτό μπορεί να έχει σοβαρές σε επίπεδο ε, σχέσεων Σαουδικής Αραβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο σχέσεων Σαουδικής Αραβίας και GCC. Ε, ε, πρέπει να υπάρξει επίκληση ώστε να ελευθερωθεί ο Ραΐφ Μπαντάουι και όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι οι οποίοι είναι κρατούμενοι επειδή εξέφρασαν τις απόψεις τους στη χώρα αυτή. Η πρόεδρο, ευχαριστούμε. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, έχετε το λόγο για να μα δώσετε περισσότερα στοιχεία. Hello, my name is Peter Γεια σα. Εκπροσωπώ το Συμβούλιο των Χωρών συνεργασία του Κόλπου στην Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Η Υπηρεσία Εξωτερική δράση παρακολουθούσε το του στην υπόθεση αυτού του κυρίου Μπαντάουι, του blogger, από όταν συνελήφθη τον Ιούνιο του 2012. Ο κ. Μπαντάουι, από ό,τι γνωρίζουμε, καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση, χίλιες, χίλιες απαγόρευση να χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης και απαγόρευση 10 ετών όσον αφορά τραξίδια, 10 ε, χρόνια μετά την αποφυλάκησή του και περίπου 230.000 ευρώ σε οικονομική αποζημίωση αυτά βγήκε από το εφετείο. Λοιπόν, οι κατηγορίες κατά του κ. Μπαντάου είναι οι εξή. Παραβίαση των Ισλαμικών αξιών, παραβίαση του Σαρία, βλασφημία, ε, λιδωρία θρησκευτικών ε, συμβόλων, χρήση στο στο διαδίκτυο, στα πλαίσια τριών φιλελευθέρων ιστοσελίδων. Μαστιγώθηκε δημοσία στις 9 Ιανουαρίου, στην Τζέντα. Ε, δέχτηκε τις 50 πρώτες βουρδουλιές. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση την ίδια μέρα έκανε ανακοίνωση. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρο, επειδή έχουμε καθυστερήσει πολύ. Η περιγραφή των γεγονότων, αν μπορείτε, να τι αφήσουμε. Ε, κοιτάξτε, η Υπηρεσία Εξωτερική δράση εξέδωσε δήλωση, ανακοίνωση την ίδια μέρα. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι σωματικές ποινές και αυτού του είδους οι ποινές είναι απαράδεκτες σε μια χώρα με ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κάλεσε τις αρχές Σαουδικής Αραβίας να μην εφαρμόσουν, να μην μας άλλο τον κύριο Μπαντάουι και στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας να εξετάσουν το δεχόμα τεθεί τέρμα στη χρήση του μαστιγώματος ως ποινή. Είναι μια ποινή που δεν συνάδει με διεθνείς αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε με τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων που έχει κυρώσει η Σαουδική Αραβία. Σε, εκτένη, σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ατύπως και επισήμως δρομολόγησε πρωτοβουλίες έναντι των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στις Βρυξέλλες και στο Ριάντ. Έκανε διαβήματα όσον αφορά τον κύριο Μπαντάουι. Η υπηρεσία μας υπογράμμισε στους συνομιλητές της Σαουδικής Αραβίας τους κινδύνους που διατρέχει η φήμη της Σαουδικής Αραβίας. Να μαυρωθεί η εικόνα της. Κυρίως και μετά τα ταγικά γεγονότα στη Γαλλία και που υπάρχει μεγάλη ευαισθησία λόγω αυτών στην Ευρώπη. Ε, και κυρίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθεί την μεγάλη δημόσια αντίδραση στην υπόθεση αυτή. Έχει γίνει εμβληματική αυτή η υπόθεση για πολύ κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύει η υπηρεσία μας ότι στο παρόν πλαίσιο οι φωνές που ζητούν μετριοπάθεια και ειρηνική δημόσια συζήτηση για διάφορα θέματα είναι κάτι που απαιτείται. Παραλλήλως, η υπόθεση του, κυρίου, του νομικού του κυρίου Μπτάμπη, του κυρίου Βαλίντ Αμπνταλ Καχύρ, επίσης είναι άκουσα ανησυχητική. Ε, στις 12 Ιανουαρίου τελικά επικυρώθη η καταδίκη του. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία που θα βρει και όλα τα διπλωματικά μέσα στη διάθεσή της τις επόμενες μέρες και όσο χρειαστεί στην περίπτωση του κυρίου Μπαντάουι. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Σοτρεβίτσιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους και το ακροατήριο ότι από σήμερα 105 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου υπέγραψαν μια επιστολή και απευθύνουν έκκληση στην ύπατη εκπρόσωπο και ζητούν κατεπηγόντως να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα όσον αφορά την υπόθεση Ραΐτ Μπαντάουι και ελπίζουμε ότι 105 υπογραφές και φωνές θα έχουν ε, κάποια επιρροή σε όλη την κατάσταση. Ευχαριστώ. Να, να σας πω Τη Είχαμε καλέσει και την πρεσβεία να παραστεί εδώ στη Σαδική Αραβία στην Ακρόαση και να πάρει το λόγο. Γιατί ήθελα, θέλαμε να μοιραστούμε μαζί τους το μήνυμα που θελήσαμε να εκπέμψουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θα συνεχίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δράση αυτή και σας παρακαλώ να κάνετε να ακουστεί η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις χώρες σας αντιστοίχως. Τώρα, εάν συμφωνείτε, να βγάλουμε μια φωτογραφία ζητώντας την απελευθέρωση του Ραΐφ Μπαντάουι μαζί με τους εκπροσώπους της Διεθνούς Αμνηστίας. Βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι θέλουν να βγουν στη φωτογραφία μαζί μας. Εδώ έξω.